we going Αρχίζουμε αγαπητοί συνάδελφοι. Καθίστε παρακαλώ. Σήμερα το απόγευμα έχουμε το προνόμιο να έχουμε μαζί μας υψηλού επίπεδου μέλη του IPCC, της Δικαιωματικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος, για να μας παρουσιάσουν τις ε, περίφημες, δυστυχώς, εκθέσεις τους για την κλιματική αλλαγή και τη γη, η νημή και την ειδική έκθεση για τους ωκεανούς, την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβελόμενο κλίμα. Και λέω δυστυχώς, γιατί ξέρουμε τι λένε οι εκθέσεις αυτές λίγο πολύ, θα μας τα παρουσιάσετε βέβαια τώρα λεπτομερώς και είναι θλιβερά αυτά που θα μάθουμε. Οπότε και εμείς οι πολιτικοί πρέπει να δράσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που βρήκατε χρόνο για να έρθετε. Ξέρω ότι ήταν δύσκολο εδώ και εβδομάδε να καταφέρουμε να βρούμε την κατάλληλη στιγμή για να μπορείτε να είσαστε και οι δύο εδώ. Σα ευχαριστούμε πάντω που ήρθατε. Τώρα, πώ θα οργανωθεί αυτή η συζήτηση. Θα οργανωθεί ω εξή. Έχουμε πρώτα απ' όλα εδώ πέρα μέλη και τη Επιτροπή Ανάπτυξη και τη Επιτροπή Αλίας. Καλώ ήρθατε. Και θα έχουμε συζήτηση λοιπόν, η οποία θα χωριστεί σε δύο τμήματα. Ε, το πρώτο τμήμα θα είναι μέχρι τις 3 και 20 περίπου και θα πρόκειται για την ειδική έκθεση του IPCC για την κλιματική αλληλεγγύη και τη γη και το δεύτερο τμήμα θα αφορά την άλλη έκθεση για τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα. Θα έχουμε 10-15 λεπτά παρουσίαση κάθε φορά και μετά catch the eye όποιος θέλει και ελπίζω να μπορέσουν όσο γίνεται περισσότεροι να πάρουν τον λόγο και μετά στο τέλος θα δώσουμε το λόγο πάλι στους προσκεκλημένους μας για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη έκθεση για την γη και το κλίμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την δυνατότητα που μας δώσετε να έρθουμε εδώ. Ε, θα κάνουμε την παρουσίαση αυτή εγώ, που είμαι ο κύριος Σκή, που είμαι ο πρόεδρος, αλλά θα είναι και ο Ζαν Φρανσουά Σουζάνα, ο οποίος ε, έχει ε, γράψει και αυτός μαζί μας την έκθεση αυτή για την κλιματική αλλαγή και τη γη. Αναφερθήκατε σε κάποια στοιχεία, θα επανέλθουμε και εμείς μετά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, η έκθεση αυτή έχει μεγάλο τίτλο και περιλαμβάνει πολλά στοιχεία και δείχνεται από πού ήρθε η έκθεση αυτή, από 7 διαφορετικές εκθέσεις για ειδικέ ε, εκθέσεις από διάφορες κυβερνήσεις που συμμετέχουν στο IPCC. Και οι διάφορες ε, προτάσεις αυτές ενσωματώθηκαν σε μία ενιαία πρόταση που έχει να κάνει με τη γη. Οι μισές από αυτές έχουν να κάνουν με την απερίμωση, την καταστροφή της γης και ένα άλλο τμήμα έχει να κάνει με τα τρόφιμα και τη δασοκομεία και τη χρήση γης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ε, μία από τις οργανώσεις των παρατηρητών που πρότεινε την ειδική έκθεση για τη γεωργία, τη χρήση γης και τη δασοκομεία. Η διάρθρωση λοιπόν της έκθεσης είναι αυτή που βλέπετε εδώ. Και θέλω να τονίσω ότι οι συντάκτες θέλαν να πρόκειται για μία ολοκληρωμένη έκθεση, να μην πρόκειται για 5, 6, 7 διαφορετικά θέματα που τα προσθέτουμε. Οπότε προσπαθήσαμε να τα ενσωματώσουμε όλα σε όλα. Οπότε ξεκινάω από την γεωργία και το πλαίσιο. Και μετά βέβαια έχουμε ε, γη, κλίμα και την αλληλοεπίδραση και μετά έχουμε τρία θέματα, τρεις στόχους, δηλαδή πώς θα αποφύγουμε την ε, απερίμωση, την καταστροφή της γης και πώς θα ασφαλίσουμε την, ε, τα τρόφιμα. Το κεφάλαιο 6 αναφέρεται στις απαντήσεις που μπορούμε να δώσουμε, τις συνέργειες που μπορούμε να προκαλέσουμε και το κεφάλαιο 7 αναφέρεται στις ε, θεσμικές συνθήκες και τις πολιτικές που μπορούν να βοηθήσουν. Πολύ σύντομα λοιπόν κάποια στατιστικά στοιχεία. 107 ήταν οι συντάκτες ε, από πέντε διαφορετικές χώρες. Το 40% ήταν οι γυναίκες και για πρώτη φορά στην ιστορία του επίσης είναι μια έκθεση η οποία έχει περισσότερους συντάκτες από αναπτυσσόμενες χώρες παρά από αναπτυγμένες χώρες. Δεν θα σας διαβάσω τα στατιστικά στοιχεία, πάντως έγινε πάρα πολλή δουλειά στην αξιολόγηση των επιστημονικών δημοσιεύσεων και μελέτη των σχολείων. Εδώ βλέπετε λοιπόν τα μηνύματα που έρχονται από την έκθεση. Πρώτα απ' όλα, ότι η γη υποβάλλεται σε πίεση από τον άνθρωπο. Αλλά επίσης η γη αποτελεί μέρος της λύσης. Υπό τον όρο βέβαια να ξέρουμε ότι η γη από μόνη της δεν πρόκειται να λύσει τα πάντα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή. Και άλλοι κλάδοι και άλλοι τομείς πρέπει να βοηθήσουν. Οπότε η γη είναι ζωτική σημασία ε, πηγή. Βασιζόμαστε σε αυτήν για τρόφιμα, για νερό, για υγεία, για ευημερία και η ανθρώπινη δραστηριότητα την επηρεάζει αρνητικά. Η κλιματική αλλαγή προσθέτει στην πίεση αυτή. Στατιστικά δεδομένα. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για 1,53 βαθμούς Κελσίου που είναι το όριο. Και η γη έχει ήδη ε, θερμανθεί πάρα πολύ 1,5 βαθμό, ε, δηλαδή παραπάνω σε σχέση με την πρώτη βιομηχανική περίοδο. Επίσης, ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία δεν είχαμε τέτοια εντατική χρήση της γης και απώλεια βιοπικιλότητας πράγματα τα οποία βέβαια έχουν αρνητικές ε, συνέπειες, η υπερεκμετάλλευση των πηγών και ο περιορισμός κάτω από τους δύο βαθμούς ε, Κελσίου, κάτι που συμφωνήθηκε στο Παρίσι, μπορεί να βοηθήσει να ε, μετριαστούν οι αρνητικές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή επί της γης. Έπειτα, οι εκπομπές. 23% των συνολικών εκπομπών είναι από τις δραστηριότητες από τη γη και πως επίσης το 44% των ε, εκπομπών μεθανίου είναι ανθρωπογενούς μορφής. Το 50% επίσης ε, αζότου που οφείλεται στη γεωργία και που δεν απορροφάται από τις καλλιέργειες. Και επίσης τα βοσκοτόπια είναι υπεύθυνα από το 1 τρίτο του, των συνολικών ε, εκπομπών οξυδίων του αζότου από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Τώρα, η επιδείνωση της κατάστασης της γης επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων. Το 1 τέταρτο επίσης της παγωμένης επιφάνειας της γης. Η χρήση της γης, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τους σπόρους και η γεωργία είναι η κύριοι τομείς και σίγουρα Ζων Φρανσουά θα σας πει περισσότερα γι' αυτό. Η κλιματική αλλαγή Επίσης επιταχύνει τον βαθμό και το μέγεθος της καταστροφής της γης και υπάρχουν επιπτώσεις και για τις ε, φυσικές πηγές, για τη ζωή των ανθρώπων αλλά και για ολόκληρες κοινωνίες. Και τέλος η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει τους ανθρώπους, τις ζωές μας, τις υποδομές. Τώρα δύο σημεία ακόμα για τα όρια της προσαρμογής και των ελεκάνων ε, αποθήκευσης ε, διοξιδίου του άνθρακα. Υπάρχουν κάποια όρια, γιατί αν χαθεί πλήρως η παραγωγικότητα, οι δυνατότητες προσαρμογής είναι πολύ μικρές, όπως επίσης και η άμβληση των επιπτώσεων περιορίζεται. Γιατί οι αποθήκες άνθρακα αλλά και τα φυτά τα οποία παροφούν διοξείδιο του άνθρακα κανονικά φτάνουν σε σημείο κορεσμού και δεν μπορούν να απορροφήσουν περισσότερο. Αυτά ήταν τα θλιβερά νέα. Τώρα, συντονισμένη δράση για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή μπορεί ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει τα θέματα της γης, της ασφάλειας τροφίμων, της πείνας, ώστε να μην υπάρχει πια πείνα. Εδώ είναι ένα διάγραμμα με διάφορες λεπτομέρειες, να σας πω τι είναι τα χρώματα. και τι μας λένε αυτά. Έχουν διάφορες απαντήσεις όσον αφορά τη γη οι συντάκτες και προσπαθούν να δούνε τι επιπτώσεις αυτές οι επιλογές μπορούν να προσφέρουν στην προσαρμογή του κλίματος, στην άμβληση των επιπτώσεων του κλίματος, στην ε, απερίμωση, στην καταστροφή της γης και στην ασφάλεια τροφίμων. Και υπάρχει ένα σκορ στο οποίο καταλήγουμε, όπου ότι είναι μπλε, είναι θετικό το αποτέλεσμα. Αν είναι πορτοκαλί, είναι αρνητικές οι συνέπειες. Και το συμπέρασμα είναι ότι πολλές από τις εναλλακτικέ λύσεις προσφέρουν πολλά ωφέλη, οπότε μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κατάσταση από όπου όλοι έχουν να κερδίσουν. Δεν φαίνεται απαραίτητα πάντα, αλλά η αγροδασοκομεία ε, και άλλα πράγματα μπορούν να έχουν πολύ θετικές συνέπειες όσον αφορά την άβληση των επιπτώσεων, κάτι για το οποίο θα σας μιλήσει ο Ζων Φρανσουά περισσότερο. Η προηγούμενη έκθεση τώρα IPCC για τον 1,5 βαθμό θέρμανση του πλανήτη αντιμετωπίστηκε με διάφορα μέτρα και διάφορες εναλλακτικές που υιοθετήθηκαν με την αποθήκευση, για παράδειγμα, άνθρακα. Και είχαμε έτσι την ευκαιρία ε, τα μηνύματα που δίναμε για τις επιλογές αυτές να μπορέσουν να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες και αποχρώσεις. Χωρίς να μιλάμε για το τι καλλιέργειες χρησιμοποιούμε ή τι μοντέλα ακριβώς ακολουθούμε, πάντως αν δεν προχωρήσουμε σε τέτοιες λύσεις, και γίνουν όλα χωρίς να έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά, δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε, αλλά πρέπει να δούμε συγκεκριμένα ε, τι κάνουμε με τις ζωοτροφές, τι άλλες επιλογές έχουμε και πού μπορούμε να έχουμε, από τι να έχουμε βιοενέργεια. Μόνο τότε μπορούμε να έχουμε ωφέλη. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό μήνυμα αυτό και περάσαμε πάρα πολύ χρόνο όταν διαπραγματευόμαστε προκειμένου να μην καταλήξουμε σε ένα έτσι χοντρικό μήνυμα που να λέει απλώ ότι η βιοενέργεια είναι κάτι κακό. Όχι, εξαρτάται πώ θα τη χρησιμοποιήσουμε και από πού θα την πάρουμε και πώς θα την πάρουμε. Επίσης αναφερθήκαμε και στο θέμα των, της των επιλογών αυτών. Τονίζουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει η μέτρηση και ο έλεγχος των αλλαγών στη χρήση γης, χρησιμοποιώντα τι σύγχρονε τεχνολογίε που μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Επίση, είναι σημαντικό να επενδύουμε στι ικανότητε των ανθρώπων, αλλά και τι θεσμικέ επίση δυνατότητε για να υπάρχει ένα σύστημα έγκαιρη προειδοποίηση που μπορεί να βοηθήσει με προβλέψεις για τα διάφορα εποχιακά φαινόμενα. Επίσης μπορούμε έτσι να βοηθήσουμε να προβλέψουμε ε, την πρόσβαση στις αγορές, τι γίνεται με την απερίμωση, στρατηγικές για την αντιμετώπιση της ή να προετοιμαστούμε για ξηρασίες, προστατεύοντας την υγεία και προσφέροντας κοινωνική προστασία. Αυτό είναι το δικό μου το κομμάτι. Πάντως το μήνυμα που βγαίνει από αυτά είναι ότι καλύτερη διαχείριση της γης μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά δεν μπορεί από μόνη της διαχείριση της γης να λύσει όλα τα προβλήματα. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον συναδελφό μου. Ευχαριστώ, Τζιμ. Σε αυτή την έκθεση έχουμε εξετάσει και το Παγκόσμιο Σύστημα Τροφίμων και τη συσχέτισή του με τις κλιματικές αλλαγές. Το Παγκόσμιο Σύστημα ε, Τροφίμων συμπεριλαμβάνει την παραγωγή, επεξεργασία, διανομή, ε, προετοιμασία και κατανάλωση των τροφίμων, ε, καθώς και τις κοινωνικο-οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή 25 με 30% του συνόλου των τροφίμων που παράγονται σπαταλώνται ή χάνονται. Οι αλλαγές στην κατανάλωση έχουν συμβάλει στο να είναι περίπου 2 δισεκατομμύρια ενήλικες υπέρβαροι ή και παχύσαρκοι. 821 εκατομμύρια άνθρωποι είναι ωστόσο ε, ε υποσυτίζονται αυτή τη στιγμή η κλιματική αλλαγή έχει ήδη επηρεάσει την ασφάλεια των τροφίμων, γιατί παρατηρούμε ότι σε πολλές περιφέρειες των χαμηλότερων ε, ε, ε, το νότιου μισφαιρίου, οι συγκομιδές κάποιων καλλιεργιών έχουν ε, μειωθεί. Αν και κάποιες άλλες ε, σοδιές, όπως α πούμε το ζαχαροκάλαμο, έχουν αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Οι κλιματικές αλλαγές έχουν ε, περιορίσει τα ποσοστά της ανάπτυξης των ζώων στην Αφρική. Επίσης υπάρχουν αυξήσεις και μειώσεις των διαφόρων νόσων. Στο μέλλον ε, γνωρίζουμε ότι μπορεί να έχουμε περαιτέρω προβλήματα με τους κινδύνους όσον αφορά τη σταθερότητα στην ε, προμήθεια τροφίμων, γιατί αυτή μάλλον θα μειωθεί, ε, ενώ το μέγεθος και η συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων που ρηγνύουν την αλυσίδα παραγωγής τροφίμων αυξάνεται. Επίσης μπορεί να μειωθεί η διατροφική ποιότητα των των διαφόρων καλλιεργειών. Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές λόγω των κλιματικών αλλαγών και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένα με 23% αύξηση στις τιμές πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο για την ανασφάλεια στα τρόφιμα. Οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι θα επηρεαστούν και περισσότερο. Επίσης, η αυξημένη ε, ε, σε θερμοκρασίες μπορεί να διευρύνουν τη μετανάστευση, ε, την εσωτερική στις χώρες, αλλά και τη διασυνοριακή μετανάστευση. Αν εξετάσουμε λοιπόν αυτό που ονομάζουμε στην ορολογία μας αυτό το χρωματικό γράφημα, όπου βλέπουμε με τη σημερινή, σημερινό επίπεδο ε, θέρμανσης, ήδη είμαστε σε σενάριο που βλέπουμε ασυνήθιστες ε, εχμές που επηρεάζουν ε, συγκεκριμένες χώρες και επηρεάζουν και τις τιμές των τροφίμων. Εάν έχουμε αύξηση θερμοκρασίας 1,5 βαθμό Κελσίου μπορεί να έχουμε σοκ διατροφικά σε διάφορες ε, περιφέρειες και εάν ξεπεραστούν οι δύο βαθμοί θερμοκρασίας μπορεί να έχουμε ρήξη στην αλυσίδα της, παροχής τροφικής αλυσίδας σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ρήξη στις μεταφορές, στην επεξεργασία και στη διανομή και οι εκπομπές δε από αυτά φτάνουν στο 21 με 37% του συνόλου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που οφείλονται σε ανθρωπογενείς ε, λόγους. Υπάρχουν όμως δυνατότητες ανταπόκρισης σε ολόκληρη αλυσίδα ε, ε, τροφίμων από την παραγωγή στην κατανάλωση και μπορεί να αναπτυχθούν και να στηρίξουν την προσαρμογή και τον μετριασμό αυτών των φαινομένων. Ναι. Έχουμε διάφορες ε, γεωργικές ε, επιλογές που μπορεί να έχουν ωφέλη ε, για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που έχουν να κάνουν με τις γέες. Το ίδιο μπορεί να σημαίνει και για τις δραστηριότητες εκτροφής ζώων όσο και για την τη γεωργία αλλά και την δασοκομεία. οι προσαρμογές, ή μάλλον οι επιλογές προσαρμογής και μετριασμού που σχετίζονται με τα τρόφιμα μπορεί να συμβάλλουν στο ε, ε, μείωση 8 με 10% των εκπομπών ε, των αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα γης μέχρι το 2050. Η διαφοροποίηση στον τρόπο διατροφής επίσης μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, όπως ας πούμε το να τρώει κανείς περισσότερα φρούτα και λαχανικά, καθώς και το να καλλιεργούνται περισσότερες ε, ε, καλλιέργειες ε, με μεγάλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. Υπάρχουν προγράμματα, συστήματα μάλλον παραγωγής, ε, με συγκεκριμένες δυνατότητες που στηρίζουν ε, την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές και το μετριασμό αυτών. Μέχρι το 2050 μπορεί έτσι να απελευθερωθούν ε, εκατομμύρια τετραγωνικά γης με ωφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και για την υγεία αλλά και να οδηγήσουν σε μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Θα ήθελα να τελειώσω δίνοντας τον επίγοντα χαρακτήρα όλων αυτών γιατί ε, αν καθυστερήσει η λήψη ε, μέτρων για την, ε, το μετριασμό των κλιματικών αλλαγών και για την προσαρμογή σε αυτά μπορεί να έχουν, μπορεί αυτό να έχει αρνητικές επιπτώσεις και για τη γη και για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και να επηρεάσει αρνητικά και με τρόπο που να μην μπορεί να αναστραφεί ορισμένα οικοσυστήματα. Η γρήγορη δράση η ταχεία δράση για τις κλιματικές αλλαγές μπορεί να οδηγήσει στην μείωση των κινδύνων για εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν ε, σε περιοχές κινδύνου. Η αναβολή δε το περικοπής των εκπομπών μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο εκατομμύρια ε, ανθρώπους. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα ακολουθήσει λοιπόν τώρα μια η διαδικασία Catch the Eye. Η πρώτη ερώτηση θα είναι προς τον Donald Τραμπ. Όχι, όχι, πλάκα κάνω. Χωρίς καμία σύγκριση βέβαια, ο πρώτος ομιλητής θα είναι ο Πίτερ Λίζε. Και βεβαίως Έχω, έχουν ζητήσει πέντε με έξι συνάδελφοι το λόγο εντωμεταξύ. Πίτερ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την παρουσίαση. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε τεράστια ευθύνη για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Το δικό μου το ερώτημα είναι πόσο δύσκολο θα είναι για τις μεταγενέστερες γενιές. Ξέρουμε ότι αν δεν δράσουμε θα έχουμε αύξηση των επιπέδων της θάλασσας κατά ένα μέτρο το 2100. Αλλά υπάρχουν και κάποια σενάρια, ίσως να μην είναι και απολύτως πιθανά, αλλά μετά από το 2100, αν αρχίσουν να λιώνουν οι κυπαγετώνες της Ιρλανδίας, θα είναι ακόμη ψηλότερη αύξηση του επίπεδου της θάλασσας. Και δεν ξέρω πόσο επιστημονικό είναι το background σε αυτό το σενάριο. Δηλαδή, αν δεν κάνουμε αυτά που πρέπει τα επόμενα 20 χρόνια, όχι μόνο η Ευρώπη, ο κόσμος, όλος ο πλανήτης, αν αποτύχουμε τελικώ, τι θα γίνει ακόμα και μετά το 2100. Εκεί νομίζω ότι είναι το πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα μόνο δύο γενεών. Ίσως είναι πρόβλημα εκατοντάδων γενεών, οπότε θέλω λίγο να καταλάβω το επιστημονικό υπόβαθρο και την πρόγνωση την επιστημονική για την περίοδο μετά το 2100. Okay, so we have César for the SND. Για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε, και ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας είπατε. Λοιπόν, γνωρίζοντας ότι υπάρχει ένας κίνδυνος, ο Λευκός Σίκος, που αποσύρθηκε από τις συμφωνίες των Παρισίων, το 20% μόνο των χωρών τηρούν τις συμφωνίες αυτές από ό,τι φαίνεται. Η Κίνα έχει το 27% των εκπομπών και δεν συμμορφώνεται. Το ΗΠΑ 13%, η Ινδία 7%, η Ρωσία το 4,6% και δεν συμμορφώνεται καμία από αυτές. Συνεπώς κυρίες και κύριοι, αν δεν κάνουμε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει εμείς μέχρι το 2050, από, 50, ε, από το 2050 και μετά, πόσο χρόνο θα έχουμε για να αντιδράσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Ρωτάω λοιπόν, πιστεύετε ότι μια πραγματική πράσινη δημοσιονομική πολιτική που να βοηθάει για τη μετάβαση μπορεί να είναι μια σωστή λύση. Renew, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεση και έχω ένα ερώτημα για το πώς βλέπουμε το θέμα συνολικά. Συζητούμε τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και κατά τη διάρκεια της παρουσίας σας ακούσαμε για την πίεση και τη διαχείριση στην γη και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και επίσης πώς μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση ε, που, θα κερδίζει, που θα κερδίζουν όλοι και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και για την ασφάλεια την επιστηστική. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθούμε για, στις προσπάθειες αυτές για να πετύχουμε τις, ε, να αντιμετωπίσουμε το κλίμα αλλά και να έχουμε ε, θετικά αποτελέσματα και για το εισόδημα των πολιτών. Κάθε γεωργικό μοντέλο έχει βεβαίως τον δικό του περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Οπότε θα ήθελα να προσπαθήσουμε να βρούμε τον βέλτιστο δυνατό τρόπο να μειώσουμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο όσο δυνατόν περισσότερο. Βέβαια, εδώ στο Κοινοβούλιο πάντα συζητούμε ποιο είναι το καλύτερο αγροτικό μοντέλο. Υπάρχουν ομάδε που λένε ε, πρέπει να έχουμε ένα πολύ παραγωγικό αγροτικό μοντέλο, γιατί έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε μεγαλύτερη, ε, μεγαλύτερο αντίκτυπο. Θα χρησιμοποιούμε λιγότερη γη για να παράξουμε τον, την ίδια ποσότητα τροφίμων και άρα μπορούμε να ε, σώσουμε κάποια κομμάτια γης για να τα διατηρήσουμε για την βιοπικιλότητα. Άλλες ομάδες λένε όχι, όχι, όλα πρέπει να είναι βιολογικά, άρα πολύ εντατική καλλιέργεια. Χρησιμοποιούμε λοιπόν ε, πολύ γη για την ίδια ποσότητα τροφίμων και αυτό μπορεί να έχει ε, αντίκτυπο. Εσείς τι πιστεύετε για αυτή τη συζήτηση και ποια μοντέλο θα πρέπει τελικώς να ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ για τους πρασίνους. Η κυρία Μπάρους, ευχαριστώ. Πολύ ε, ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Πρέπει να πω ότι δεν έχω διαβάσει πλήρω την ε, ε, έκθεσή σας. Διάβασα μόνο την περίληψη για τους χαράσοντες πολιτικοί και δεν μπορώ να πω ότι είδα κάποια σαφή παρέμβαση για την διάβρωση της γης που, εν, που επιτείνεται από κάποια είδη ε, γεωργίας για την αποθήκευση άνθρακα. Θα ήθελα να μου πείτε αν μέσα στην έκθεση υπάρχουν σχετικά στοιχεία. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάζελκαμπ για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Η έκθεση σας δείχνει ότι πρέπει να συζητήσουμε πολύ περισσότερο για τα τρόφιμα όταν μιλούμε για την κλιματική αλλαγή. Ένα μήνυμα που ελπίζω ότι και οι συνάδελφοι εδώ στην Επιτροπή ΕΜΒΗ και στη ΔΕΒΕ ε, θα λάβουν σοβαρά υπόψη τους, αλλά και στην Κομισιόν. Μιλάτε για διατροφικές αλλαγές, για αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, για να αποφύγουμε την οικολογική και περιβαλλοντική κατάρρευση και μιλάτε για διάφορες δράσεις που μπορούν να βοηθήσουν προς αυτό. Μπορείτε να μας πείτε κάποιες προτεραιότητες για τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να γίνουν αυτές οι αλλαγές στις διατροφικές μας συνήθειες. Και δεύτερο ερώτημα που θέλω να σας θέσω. Στην έκθεση μιλάτε για την ανάγκη του να μεταφερθούμε σε, μια πιο βιώσιμη, διατροφή, σε πιο βιώσιμες διατροφικές συνήθειες. Γιατί εκεί μιλούμε για, τις, ε, για πολύ μεγάλες ε, εκπομπές σε σχέση με το σύνολο των, του τομέα των μεταφορών. Η Γεωργία κυρίως ε, η παραγωγή ε, ε, ζωοτροφών και γαλακτοκομικών έχει μεγάλο μερίδιο στις παγκόσμιες εκπομπές αερίων. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα και πώς θα μπορούσαμε να αναδιαρθρώσουμε τις εμπορικές και γεωργικές πολιτικές μας ως προς αυτό. Ελπίζω να μπορείτε να μας πείτε και κάτι για τις τεράστιες ε, ε, γεωργές επιδοτήσεις και για την πρόθεση της όλης πολιτικής ε, κατανάλωσης κρέατος και γαλακτοκομικών. Η κυρία Νταλή για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τους ειδικού που είναι εδώ, τους εμπειρογνώμονες και που μας παρουσίασαν τα ευρήματα της έκθεσής τους. Συχνά μιλούμε για τις μελλοντικέ γενιές, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας. Πολλοί νομίζω ήδη αισθανόμαστε τον αντίκτυπο σήμερα και από ό,τι καταλαβαίνουμε και από την έκθεση. Αν δεν κάνουμε επίγοντα, αν δεν λάβουμε επίγοντα μέτρα, όπως είπαν και οι εμπειρογνώμονες, τα αποτελέσματα θα συνεχίσουμε να τα νιώθουμε όχι μόνο εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, αλλά και ε, οι επόμενες γενιές. Είδαμε ότι πρέπει να, γίνει, να υπάρξουν άμεσες δράσεις, επίγουσες, αν θέλουμε να αποφύγουμε τον αρνητικό αντίκτυπο. Και είναι πιθανό, είναι δυνατό οι εμπειρογνώμονες να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες για το τι σημαίνει επίγουσα δράση. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές διατρέχουμε, συζητούμε αυτές τις εκθέσεις, ακούμε πολύ ωραία λόγια και εδώ στο κοινοβούλιο, αλλά όταν περνάμε σε απτά μέτρα και τι μπορούμε να κάνουμε μέσω της νομοθεσίας και μέσω επιγουσών δράσεων, τότε αρχίσουμε να κάνουμε φιλοσοφικές συζητήσεις για το τι θα πρέπει να είναι μια επίγουσα δράση. Αν θέλουμε όντως να τηρήσουμε το 1,5, τον 1,5 βαθμό αύξησης θερμοκρασίας και να τον αντιμετωπίσουμε, θα πρέπει πρακτικά να μας πούν οι επιστήμονες αν θεωρούν ότι τα μέτρα που έχουν υπάρξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα μέτρα που προτείνονται για να ληφθούν αν θεωρούνται όντω επίγουσα δράση ή αν πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο. Και αν ναι, ποιο είναι αυτό το περισσότερο, ποια είναι αυτή η επίγουσα δράση πρακτικά που μπορεί να υπάρξει. Ευχαριστώ. Για το ΕΛΚ, Νόβακ. Ευχαριστώ. Αναρωτιέμαι κατά πόσο μπορούμε πραγματικά να καταφέρουμε κάτι αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Ακούμε όλο και περισσότερα μαγαζιά, δημιουργούνται περισσότερα σούπερ μάρκετ, καταναλώνουμε όλο και περισσότερα. Η γεωργία δεν είναι υπεύθυνοι για την βιοπικιλότητα. Εμείς, ο τρόπος με τον οποίο εμείς ζούμε είναι υπεύθυνο, ο τρόπος που καταναλώνουμε. Έχουμε περισσότερα αυτοκίνητα, θέλουμε περισσότερους δρόμους. Έχουμε καταστρέψει πάρα πολλά είδη, έχουμε καταστρέψει πολλά. Και αναρωτιέμαι κατά πόσο όλα αυτά τα μέτρα θα μας επέτρεπαν πραγματικά να επηρεάσουμε την κλιματική αλλαγή ή μήπως πρέπει πραγματικά να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας. Ευχαριστώ. Κλείνει ο κατάλογος, γιατί έχουμε πολλούς. Ρινιού Μαρτίν Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ για την παρουσίαση. Είναι αλλιώς να τα ακούει κανείς και να τα διαβάζει. Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία έχει να κάνει με την ενέργεια και θέλω να ακούσω την διενέργεια. Ε, δεδομένων των ενστάσεων. Θα ήθελα να ξέρω περισσότερα. Εσείς πώς βλέπετε την ευρωπαϊκή πολιτική προσφέρει κάτι θετικό και αποφεύγει τα αρνητικά και τι συστάσεις θα είχατε να κάνετε ε, για το πώς θα πρέπει να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, επειδή πραγματικά πρόκειται για μια παγκόσμια δράση. Ήθελα να ξέρω εσείς στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα βλέπετε να υπάρχει χώρος ώστε να έχουμε πιο πράσινα δημοσιονομικά. Θα μπορούσε αυτό να βοηθήσει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Κλάους Πούχνερ, πράσινη. Ευχαριστώ. Δύο σύντομες παρατηρήσεις. Η πρώτη. Ακούστηκε πριν λίγο ότι η βιολογική καλλιέργεια χρησιμοποιεί πάρα πολλές μεγάλες γέες για την παραγωγή τροφίμων και καλό ήταν, είναι να γίνεται πιο εντατική καλλιέργεια. Αυτό δεν είναι σωστό. Το ξέρουμε δυστυχώς από ατυχή πειράματα σε μικρές ε, περιοχές που σημαίνουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα ανά εκτάριο για την παραγωγή τροφίμων. Και επίσης η κτηνοτροφία, κυρίως για τις αγελάδες. Πρέπει να δούμε εκεί τι γίνεται με τις ζωοτροφές. Ανάλογα το, με ανάλογα τη ζωοτροφή παράγονται περισσότερα ή λιγότερα, περισσότερες ή λιγότερες εκπομπές μεθανίου. Το μεθάνιο είναι πολύ μικρότερο όμω ε, οι εκπομπέ μεθανίου από τι αγελάδε και την κτηνοτροφία είναι πολύ, πολύ μικρότερε από, από τι εκπομπέ μεθανίου σε σχέση με την εντατική καλλιέργεια ή την βιολογική καλλιέργεια. Για την ECR. Κύριε Πρόεδρε, η κυρία Ζαλεύσκα, χάρηκα πολύ που άκουσα τις παρουσιάσεις. Ήταν σύντομες βέβαια, έτσι έπρεπε φαντάζομαι, αλλά υποθέτω ότι οι ομιλητές ε, περιμένουν πολλά ερωτήματα ε, των οποίων η απάντηση δεν βρίσκεται εντός της έκθεσης. Με όλη αυτή την έρευνα που έχει γίνει, ε, δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει η φράση «κάτι πρέπει να γίνει». Είναι λίγο ασαφές, είναι λίγο φλού αυτό. Χρειαζόμαστε ε, επιλογές που να μπορούμε να ακολουθήσουμε. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούμε ότι η, ε, τα επιστημονικά στοιχεία έρχονται και η έρευνα έρχεται από αναπτυσσόμενες χώρες. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε ποιο είναι το συμπέρασμα από αυτές τις εκθέσεις και τις έρευνες. Και τέλος, ίσως θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε αυτοί που κάνουν αυτές τις μελέτες, που αναλαμβάνουν αυτές τις έρευνες, πώς επιλέγονται. Πώς ορίζεται δηλαδή ποιος θα κάνει την έρευνα. Λοιπόν, για την ΚΟΙ ο κύριος Κόκαλης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την IPCC που έθεσε την, ε, ε, το πρότυπο για την ε, πολιτική με βάση τα επιστημονικά στοιχεία και ευχαριστώ και τους ε, παρουσιάζονται τις εκθέσεις. Καταρχάς, μιλούσαμε για την διευκόλυνση των διαφόρων ε, ε, επιλογών που έχουμε, όπως το σενάριο 2,6 και μας είπατε ποια είναι η δική σας άποψη για το Green Deal της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα ψηφίσουμε τον επόμενο μήνα και ελπίζουμε ότι και στις ΕΠΑ μετά τις εκλογές του 2020 του Νοεμβρίου αν έχουν και αυτοί ένα νέο Green Deal, να ε, επανέλθουν στη Συμφωνία των, ε, του Παρισιού. Οπότε, στο μέλλον θα μπορέσετε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για το, για το όλο και αυξανόμενο α, ε, κόστος των εκπομπών του θερμοκηπίου. Και επίσης, το μέλλον της IPCC ποιο είναι, η επόμενη αποστολή σας δηλαδή ποια είναι, να παρέχετε μικρότερες, ε, μικρότερο φάσμα ας πούμε, επιλογών στην, ε, ε, στις εκθέσεις σας περνάτε περισσότερο από τις φυσικές επιστήμες, τις οικονομικές, να παρέχετε αναλύσεις κόστους ωφέλους. Αυτές είναι οι δικές μου ερωτήσεις. Και η πρότασή μου, αν μου επιτρέπετε να την κάνω, είναι να αλλάξει το ανθρωπογενές και να γίνει ανθρωποκτόνο. Ευχαριστώ να κάνετε μία έκθεση πρωτοβουλίας για το Renew. Ο κύριος Στεφανούτα. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τους δύο εμπειρογνώμονες για τις ε, τόσο ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους. Το περιοδικό Economist παρουσιάζει κάποιες τεχνικές και επιστημονικές λύσεις για να αντιμετωπιστεί το μεθάνιο πρόκειται για λύσεις 20 φορές ε, παραπάνω από ό,τι έχουμε μέχρι τώρα από τον Economist. Το αποτέλεσμα πάντως των ερευνών δείχνει θα μπορούσαμε μέχρι και 80% να μειώσουμε τις εκπομπές μεθονίου αν ε, δεν ε, εκτρέφαμε βοηθή. Ναι, μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό και σίγουρα τις γνωρίζετε όλες αυτές τις προτάσεις και ιδέες. Πάντως οι παρουσιάσεις σας, πρέπει να πω, είναι πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά έχουμε την εντύπωση ότι ζούμε σε συλλογική κατάθλιψη και ξεχνάμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε έρευνες ακριβώς για να μπορέσουμε να βγούμε από το αδιέξοδο. Πολλές φορές έχουμε ξεπεράσει τέτοιες δυσκολίες στην ιστορία της ανθρωπότητας, οπότε θα ήθελα να μας προτείνετε τεχνικές λύσεις. Ευχαριστώ. Τι της πράσινη. Η κυρία Μέτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίαση, η οποία υπογραμμίζει πόσο πολύ επίγει να προστατεύσουμε ε, το έδαφο όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε τρίτες χώρες. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το μήνυμα να το παίρνει και να το παίρνει σοβαρά και να φροντίσει για την προστασία του εδάφου όσο γίνεται πιο γρήγορα. Θέλω να ρωτήσω για τη Γεωργία συγκεκριμένα. Η έκθεση του EPCC λέει ότι τα χημικά επηρεάζουν επίσης τη γη και οδηγούν σε περισσότερες εκπομπές του θερμοκηπίου. Το συμπέρασμά σας όμως δεν λέει συγκεκριμένα ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να τρώμε και να παράγουμε όπως κάναμε μέχρι τώρα. Ούτε αναφέρονται συγκεκριμένες μελέτες που μιλάνε για τις χαμένες ευκαιρίες αποθήκευσης ε, άνθρακα. Όταν λοιπόν μετράμε τις εκπομπές εξαιτία της γεωργίας ή της χρήσης γης, δεν πρέπει να ρωτάμε ένα τρακτέρ μόνο πόσο εκπέμπει, αλλά επίσης πόσο θα μπορούσαμε να αποθηκεύσουμε ένα διαφορετικό σύστημα παραγωγής τροφίμων. Εσείς ε, λέτε ότι αν ε, τρώμε διαφορετικά μπορούμε να προστατεύσουμε το 75% της γης που πηγαίνει τώρα στη Γεωργία. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτή η γη τότε για να ε, διορθωθεί η ζημιά που έχει γίνει στο οικοσύστημα. Ωραία, τώρα έχετε 10 λεπτά για να απαντήσετε στις πολυάριθμες ερωτήσεις. Φοβάμαι, μια που έκθεσή μας είναι 1200 σελίδες, θα σας απογοητεύσουμε σε έναν βαθμό τουλάχιστον, δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω πάντως. Και ο Ζαν Φρανσουά θα απαντήσει σε άλλες αυτές που έχουν να κάνουν περισσότερο με τη Γεωργία και τα τρόφιμα. Ρωτήσατε για το ίδιο το έργο του IPCC, ε, ποιο είναι ο σκοπός Πρέπει να σας πω το ότι το IPCC δεν κάνει έρευνα, αλλά αξιολογεί την έρευνα που έχουν κάνει άλλοι και δημιουργεί και μία σύνθεση. Οι συντάκτες ορίζονται από τις κυβερνήσεις τους και από τις οργανώσεις παρατηρητών, μεταξύ άλλων και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρατηρητής. Και υπάρχει ένας κατάλογος λοιπόν και η επιστημονική ηγεσία του ΕΠΣΣ, το γραφείο, το προεδρείο κατά κάποιο τρόπο, τους επιλέγει. Συνήθως έχουμε έξι φορές περισσότερες προτάσεις από αυτούς που τελικά επιλέγουμε και προσπαθούμε να έχουμε μια ισορροπία, ανα αναγεωγραφική κατανομή κλπ. Αναπτυσσόμενες, αναπτυγμένες χώρες κλπ. Ο κύκλος αυτό το EPCC, δεν έχει ολοκληρωθεί. Η ομάδα ε, για την πρώτη ομάδα το 2021 θα έχει ολοκληρώσει τις εκθέσεις και εκεί θα απαντώνται πολλές από τις ερωτήσεις σας. Οπότε, εγώ είμαι υπεύθυνο για την ομάδα εργασία 3 που αναφέρεται στο μετριασμό και είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα ολόκληρο κεφάλαιο για την ανθρώπινη συμπεριφορά, την ανθρώπινη κατανάλωση. Προσπαθούμε δηλαδή να καινοτομήσουμε εδώ. Τώρα για τις ερωτήσεις σας. ρωτήσατε, χρειάζεται φορολόγηση του άνθρακα. Το άλλο όμως για το IPCC που πρέπει να σας πω και που μας λένε οι κυβερνήσεις είναι ότι εμείς δεν προτείνουμε πολιτικές, ούτε κάνουμε συστάσεις. Ό,τι λέμε πρέπει να τα λέμε με διαφορετικό τρόπο, να τα διατυπώνουμε διαφορετικά, όχι σαν συστάσεις ή προτάσεις πολιτικής. Μπορούμε να πούμε ποια μέσα θα βοηθούσαν περισσότερο για να πετύχουμε τον ένα ή τον άλλο στόχο. Οπότε η φορολόγηση μπορεί να αποτελεί μέρος, αλλά θα υπάρχουν και άλλες επιλογές. Ρωτήσατε για το τι μπορούμε να κάνουμε βραχυπρόθεσμα, επειδή επήγει το θέμα. Ακόμα και δεν έχετε χρόνο να διαβάσετε ολόκληρη την έκθεση, διαβάστε το τμήμα Δέλτα που έχει τον τίτλο «Βραχυπρόθεσμες δράσεις». Εκεί είναι που μιλάμε για το επίγον του θέματος και τι θα μπορούσε να γίνει για να προχωρήσουμε στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή. Αναφέρονται μέτρα όπως ε, μεταφορά γνώσης, τεχνολογίας, ε, οικονομικοί μηχανισμοί Δεν είναι σε 10 λεπτά βέβαια που μπορεί κανείς να μιλήσει για όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Τώρα το τελευταίο που θα ήθελα να πω πριν δώσω το λόγο στο Ζω Φροσουά είναι ότι υπήρξε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στην έκθεση ότι οι λύσεις πρέπει να κοπούν και ραφτούν στα μέτρα των τοπικών κοινοτήτων και των τοπικών συνθήκων. Δηλαδή μια λύση που είναι καλή στην Ευρώπη μπορεί να μην είναι καλή κάπου αλλού, στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική. Ακόμα και στα βασικά κεφάλαια ε, το λέμε αυτό. Οπότε εντοπίζουμε διαφορετικά συστήματα γεωργίας που μπορούν να συνεισφέρουν στην επιτευξή των στόχων του μετριασμού, της προσαρμογής, την αποφυγή της καταστροφής της γης κτλ. Δεν μπορείς να πιστεύεις ότι μία λύση είναι καλή για όλους. Το ίδιο ισχύει και για τη διατροφή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι καλό είναι να είναι όλοι ε, χορτοφάγοι ή αυστηρά χορτοφάγοι, vegan. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές διατροφές που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Θα δώσω το λόγο τώρα στο Ζαν Φρανσουά, αλλά να ξέρετε ότι πολλές από τις ερωτήσεις σας έχουν τις απαντήσεις στην έκθεσή μας αλλά δεν είναι δυνατόν μέσα σε 10 λεπτά να σας τις παρουσιάσω όλες. Ευχαριστώ. Αυτό το οποίο εκπλήσει με τα αποτελέσματα της έκθεσής μας είναι ότι βλέπουμε ότι πολλές από τις προτινόμενες επιλογές παρουσιάζουν σημαντικά ωφέλη. Και αυτό είναι σημαντικό σαν μήνυμα για την πολιτική και τους πολιτικούς. Γιατί στη Γεωργία, για παράδειγμα, βλέπουμε πολιτικές για την προμήθεια τροφίμων ή για τα ύδατα, για την βιοπικιλότητα, για το κλίμα. Αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον πάντως στα ευρήματα της έκθεσης είναι ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες επιλογές από τις οποίες ε, έχουμε ωφέλη για όλες τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με το κλίμα. Το θέμα είναι πώς θα στηρίξουμε την αλλαγή για να υλοποιηθούν αυτές οι επιλογές. Πιο συγκεκριμένα, πράγματι κάποιες από τις επιλογές, για παράδειγμα μείωση της ε, διάβρωσης της γης και άρα της καταστροφής της, ευθυγραμμίζεται με το θέμα του διοξιδίου του άνθρακα, δηλαδή να έχουμε ε, περισσότερες οργανικές ε, ουσίες και θα μπορούσαμε έτσι να έχουμε ωφέλη για πολλές πλευρές του προβλήματος. Πράγματι, υπάρχει κάποια ένταση. Τι μπορείς να κάνεις με, από τη μια μεριά, πιο εντατική καλλιέργεια σε πιο μικρές περιοχές και από την άλλη μεριά να προστατεύσεις τη βιοπικιλότητα αλλού. Πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε λιγότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από το σύστημα παραγωγής τροφίμων. Πάντως βλέπουμε ότι ακόμα και αν ξεκινήσουμε από τετατικά συστήματα παραγωγής, υπάρχουν επιλογές για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προστασία της γης, αναφέρονται στην έκθεσή μας και μπορούν να συνδυαστούν και μεταξύ τους. Αν επίσης συνδυάσετε ε, διαφορετικές λύσεις για την προμήθεια και την ζήτηση, μόνο ωφέλη έχετε. Και όσον αφορά τους τρόπους διατροφής, σίγουρα υπάρχουν ε, συνέργειες. Το σημείο κίνησης εδώ στην Ευρώπη είναι ότι έχουμε την τάση να καταναλώνουμε υπερβολικά πολλά ζωικά προϊόντα. Σίγουρα παραπάνω από τις κατευθυντήριες γραμμές που υπάρχουν όσον αφορά την κατανάλωση κρέατος. Οπότε εκεί θα μπορούσαμε να είχαμε ωφέλη από την αλλαγή της διατροφής. Αλλά η έκθεσή μας δείχνει το τοπίο των εναλλακτικών και των ωφελών. Τίποτα άλλο. Επιτρέψτε μου να προσθέσω μία παρατήρηση ακόμα μετά από αυτά που είπε ο Ζαν Φρανσουά και θα μπω λίγο στα χωράφια του. Το θέμα της δίκαιας μετάβασης είναι κάτι το οποίο με νοιάζει πολύ γιατί εγώ στη Σκωτία ασχολήθηκα στην κυβέρνηση εκεί με το θέμα αυτό και όταν συζητάμε με τους γεωργούς νιώθουν απειλή από τις δράσεις για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι χρειαζόμαστε οικονομικά κίνητρα, ώστε οι αγρότες και άλλοι να έχουν κίνητρα, ώστε να διαχειριστούν καλά ε, το έδαφος, τη γη και να ξέρουν ότι η γονιμότητα του εδάφους θα αυξηθεί. Αυτή τη στιγμή δεν τα μετράμε καλά όλα αυτά, όλους αυτούς τους παράγοντες. Αν το κάνουμε και δώσουμε και κίνητρα, θα βοηθήσουμε πάρα πολύ ώστε οι αγρότες να συμπλέψουν με τις προσπάθειές μας ε, για τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος. Σας ευχαριστώ. Θέσατε και ερωτήσεις για την ε, εισαγόμενη ε, αποδάσωση, αποψήλωση των δασών. Είναι αλήθεια ότι αν οι δικές μας πολιτικές εφαρμοστούν μόνο η γεωργική παραγωγή στην Ευρώπη, ε, τότε προφανώς θα έχουμε ζητήματα με το αποτύπωμα των Ευρωπαίων κρατών όσον αφορά την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου που εισαγόμενα τρόφιμα και εισαγόμενες ε, ίνες και πρωτεΐνες. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε όταν ε, προβληματιζόμαστε για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με τα θέματα γεωργίας και τροφίμων. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προχωρήσουμε στη δεύτερη ε, συνεδρία για ε, τον ωκεανούς. Πριν να περάσουμε όμως αυτό θα κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Πρώτον, ότι ο τύπος ε, ότι μάλλον θα ε, κυκλοφορήσει ένα ανακοινωθέν τύπου που θα μπει στο site μας και επίσης έχουμε ψηφοφορίες στις 4. Μην ξεχάσετε λοιπόν τις κάρτες ψηφοφορίας σας. Και τώρα έχετε πάλι το λόγο για την δεύτερη έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ονομάζομαι Hans Gertner και είμαι συνσυντάκτης της ομάδας ε, της IPCC Παριθμών 2 που ασχολούμαστε με τις δυνατότητες προσαρμογής και τα ευάλωτα ε, σημεία. Και με χαρά θα σας παρουσιάσω την έκθεσή μας για τους ωκεανούς και την κρυοσφαίρα βάλαμε αυτό το σύντομο τίτλο. Αυτή η έκθεση εκπονήθηκε από την ομάδα εργασίας 1 και 2 της ε, IPCC, γιατί η ομάδα εργασίας 3 δεν είχε τόσες επιλογές και αυτό επιβεβαιώθηκε και στη διάρκεια της αξιολόγησης, γιατί δεν είχαν πολλές δυνατότητες να ασχοληθούν με αυτά τα συστήματα και θα κάνουμε μια συνολική ε, εποπτική έκθεση στην ε, βασική έκθεση. Έχω αφαιρέσει τις στατιστικές από την έκθεση, αλλά είναι παρόμοια με αυτά που ακούσατε για τη γη όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ φύλων και περιφερειών. Και υπάρχει ένα γενικό μήνυμα που προέρχεται από αυτά τα συστήματα, για να το τονίσω, ότι οι άνθρωποι κατοικούν γύρω στο 20% του πλανήτη, αλλά σε αυτή την έκθεση μιλάμε για το επόμενο 80% που είναι η, η, και η, η κρυοσφαίρα. Εδώ και δεκαετίες μιλάμε για την ε, θέρμαση, για τις κλειδηματικές αλλαγές και θα δούμε ποιες είναι οι συνέπειες για την ανθρωπότητα και την φύση, οι οποίες είναι συντριπτικές και ε, ε, πολύ έντονες και ορισμένες έχουν ήδη συμβεί. Το θέμα ακολουθεί και τη δομή των κεφαλαίων. Θα μιλήσουμε ακολουθώντας τη ροή του νερού από τα ψηλά βουνά, τις πολικές περιοχές προς τους ωκεανούς. Και θα δούμε τι σημαίνει αυτό και ποιες είναι οι, εποπτείες των, οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στα διάφορα οικοσυστήματα. Το ένα κεφάλαιο έχει να κάνει με τα, τις οροσυρές και έχουμε την εξή δήλωση. Τα μικρά, ε, οι μικροί παγετώνες που υπάρχουν στην Ευρώπη, την Ανατολική Αφρική, τις τροπικές Άνδες και την Ινδονησία θα χάσουν πάνω από το 80% της μάζας πάγου μέχρι το 2100 εάν συνεχίσουν να αυξάνονται εντόνως οι κομπές. Καθώς οι πακετώνες λιώνουν και, και συρρυκνώνεται η κάλυψη από χιόνι, θα ανεβούν προς τα πάνω, προς τα υψηλότερα μέρη των βουνών, τα διάφορα φυτά και ζώα τα οποία ζουν χαμηλότερα αυτή τη στιγμή. Ένα σύνολο 670 εκατομμυρίων ανθρώπων ε, ζουν στις ε, περιοχές αυτές των οροσυρών και τώρα αυτοί εκτίθενται σε κινδύνους και αλλαγές όσον αφορά τη διαθεσιμότητα νερού. Η υποχώρηση της κρυοσφαίρας θα συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά τις διάφορες δραστηριότητες αναψυχής, τον τουρισμό και τις ε, πολιτιστικές αυτές δραστηριότητες. Θα περιοριστούν όλες αυτές οι δραστηριότητες λοιπόν στα ψηλά βουνά λιγότερο σκι λοιπόν στις Άλπες για πολλούς από εσά. Δεύτερο ε, θέμα είναι οι πολικές περιοχές και οι πολικοί ωκεανοί. Και εδώ έχουμε την εξή σύνοψη, ότι δηλαδή ο πάγος στην ακτική θάλασσα περιορίζεται κάθε μήνα του χρόνου και γίνεται και πιο λεπτός. Ο Αρκτικός ωκεανός δεν θα έχει πια ε, πάγο στη θάλασσα το Σεπτέμβριο και αν η αύξηση της θερμοκρασίας είναι 2 βαθμοί, αυτό θα συμβαίνει ένα στα τρία χρόνια. Βλέπετε ποια διαφορά κάνει λοιπόν όταν μιλάμε για 1,5 βαθμό αύξηση θερμοκρασίας ή για 2 βαθμούς. Επίσης οι μόνιμοι παγετώνες ε, ε, λιώνουν και αυτό μπορεί να προσθέσει περισσότερο αέριο του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Εάν οι εκπομπές αρχίσουν να αυξάνονται εντόνως, γύρω το 70% των μόνιμων παγετώνων θα χαθεί. Οι άνθρωποι που ζουν στην Αρκτική, ιδιαίτερα οι αυτόχθονες, ήδη επηρεάζονται από τις κλιματικές αλλαγές και προσαρμόζονται στην εποχικότητα και την ασφάλεια των συνθηκών στη γη, στον πάγο και στο χιόνι. Η επιτυχία τους εξαρτάται από τη χρηματοδότηση, τις δυνατότητες και τη θεσμική στήριξη. Περνάμε τώρα στον ωκεανό εν γέννη και θα μιλήσουμε και για την... Ε, κλιματικές αλλαγές σε σχέση με το τι σημαίνουν αυτές για τη θαλάσσια ζωή. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι μέχρι σήμερα ο κενό καλύπτει το 90% της υπερβολικής θέρμανσης που ε, δημιουργείται στο κλιματικό σύστημα και αυτό θα συνεχιστεί. Η θέρμανση των ωκεανών ε, περιορίζει την ανάμειξη ανάμεσα στα διάφορα στρώματα νερού και γι' αυτό περιορίζει και την παροχή οξυγόνου και, και... και στοιχείων διατροφής για τη θαλάσσια ζωή. Ε, τα θερμά θαλάσσια ρεύματα και κύματα γίνονται πιο συχνά και πιο έντονα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις περιοχές όπου υπάρχουν κοράλια. Ε, το 20 με 30% των εκπομπών θα συνεχιστεί και θα αυξάνεται εφόσον συνεχίζεται η θέρμανση του πλανήτη. Επίσης αξιολογούμε το κίνδυνο για τα οικοσυστήματα στις ε, θαλάσσιες περιοχές, στον ωκεανό αλλά και στις ακτές και έχουμε ε, δει και το ε, γράφημα που πηγαίνει από το κίτρινο μέχρι το βαθύ μόβ. Θα δείτε εδώ ότι οι διαφορές είναι μεγάλες ανάμεσα, ανάμεσα στο 1,5 και στον, στους 2 βαθμούς στα ε, στους κοριαλιογενείς υφάλους η, ε, γίνεται αισθητή ήδη. Και εδώ βλέπουμε την πρόσφατη αύξηση της θερμοκρασίας που είναι κάτω από το 1, 1 βαθμό μέχρι στιγμής. Αυτό που βλέπουμε εδώ λοιπόν είναι ότι οι κοραλογενή ύφαλοι σε θερμό νερό ήδη κινδυνεύουν πάρα πολύ. Ακόμα και με 1,5 βαθμό αύξηση δημοκρασία θα χάσουμε το 70 με το 90% των κοραλογενών ε, συστημάτων. Ε, θα χαθεί επίσης η αλληλεία μικρής κλίμακας ε, καθώς και η ε, προφύλαξη των ακτών. Εάν καταφέρουμε όμως να μείνουμε στον 1,5 βαθμό αύξησης θερμοκρασίας αντί για 2, πολλά από τα άλλα συστήματα δεν θα μετακινηθούν προς την, προς την περιοχή υψηλού κινδύνου. Δηλαδή, τα λιβάδια με φύκια, οι βραχώδεις ακτές, τα έλι με αλατισμένο νερό, ε, τα κοράλια που ζουν σε κρύο νερό δεν θα κινδυνεύουν ούτε τα δέλτα των ποταμών, ούτε και οι αμμώδεις ε, ακτές. Υπάρχουν όμως επιπτώσεις ε, που επηρεάζουν τη θαλάσσια ζωή, ιδιαίτερα αν δούμε τον περιορισμό της αύξησης ε, της ε, θερμοκρασίας των ωκεανών. Και εδώ βλέπουμε τι θα σημαίνει αυτό για τα λιεύματα. Τα καφέ χρώματα, τώρα εδώ δεν φαίνονται πολύ καλά τα χρώματα σε αυτή τη διαφάνεια, αλλά πάντως τα καφεδί δείχνουν εκεί που θα έχουμε μειώσεις, ενώ τα ε, γαλανά θα δείχνουν εκεί που θα είναι περισσότερη η αύξηση τα αλλιεύματα και δηλαδή τα, οι αλλιευτικοί πόροι ε, θα μετακινηθούν και οι τάσεις αυτές τονίζονται ακόμα περισσότερο όσο περισσότερο αυξάνεται η θερμοκρασία. Το 1,5 βαθμός ο φιλόδοξος στόχος του Παρισιού είναι αυτός που πρέπει, στον οποίο θα πρέπει να επιμείνουμε και να παραμείνουμε. οι αλληλευτικοί πόροι θα ανακατανεμηθούν και αυτό θα σημάνει πολιτικές συζητήσεις ανάμεσα στις χώρες αλλά και προκλήσεις για τις τοπικές κοινότητες. Ας συνοψίσουμε λοιπόν αυτά τα οποία μπορούμε να πούμε σε σχέση με τη θαλάσσια ζωή. Αυτή ειδικεύεται και εξαρτάται από περιορισμένες αλλαγές θερμοκρασίες. Οι αλλαγές στους ωκεανούς σημαίνει μετακίνηση των ε, πληθυσμών των αλλιευμάτων και στο μέλλον κάποιες περιοχές θα δουν μείωση των αλευτικών πόρων ενώ σε άλλες θα υπάρξει αύξηση. Οι κοινότητες θα εξαρτώνται από αλληλεύματα ε, ε, αλλιεύματα αλλά εάν μειωθούν άλλου είδους πιέσεις όπως η ρήπανση, αυτό μπορεί να βοηθήσει στη θαλάσσια ζωή και μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των ε, κλιματικών αλλαγών. Τώρα ας δούμε και ένα άλλο θέμα που αναφέρεται και ήδη στη συζήτηση και αυτό αφορά την ε, αύξηση των επιπέδων ε, της θάλασσας. Εδώ έχουμε διάφορα μοντέλα όπου έχει υπάρξει μετριασμό. αυτό είναι το θαλασσί που βλέπετε σε αυτά τα γραφήματα, ενώ εάν οι εκπομπές αυξηθούν περισσότερο, ε, έχουμε το κόκκινο ε, Έχουμε το κόκκινο χρώμα. Εδώ βλέπετε τι θα γίνει εάν λιώσουν οι παγετώνες στα ψηλά βουνά, εάν περιοριστεί ο νημόνιμοι παγετώνες στην Αρκτική και στην Ανταρκτική. Βλέπουμε δηλαδή την αύξηση το, την, την ύψωση του επίπεδου της θάλασσας μέχρι το τέλος του αιώνα βλέπουμε ότι θα φτάσουμε σε αύξηση τριών μέτρων και αυτές οι εξελίξεις θα συνεχιστούν μέχρι το 2000 400 όπου θα φτάσουμε σε ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις στο ύψος του επίπεδου της θάλασσας. Εάν περιοριστούν οι υπομπές, μπορούμε να σταθεροποιήσουμε την αύξηση του επίπεδου της θάλασσας κάτω από το 1 μέτρο μέχρι το 2300 και να φτάσουμε σε κάποιο είδος ε, σταθεροποίησης. Σύμφωνα με τις γνώσεις που έχουμε μέχρι στιγμής έχουμε επιλογές στο να μείνουμε κάτω από το 1 μέτρο ή στο να περάσουμε στην αύξηση κατά πολλά μέτρα. Αν συνοψίσουμε λοιπόν, ε, οι παγετώνες χάνουν όγκο, ε, συνεχίζει η τήξη, 680 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε ε, ακτές οι οποίες κινδυνεύουν, 65 εκατομμύρια σε μικρά νησιωτικά κράτη και θα επηρεαστούν ανάλογα με τη συνέχιση των εκπομπών ή όχι. Στη διάρκεια του 20ου αιώνα το παγκόσμιο μέσος όρος ε, του ύψους της θάλασσας αυξήθηκε κατά 15 περίπου εκατοστά, αυτή τη στιγμή η αύξηση του επίπεδου της θάλασσας ε, γίνεται σε, με διπλάσιο ρυθμό από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό σημαίνει ότι πέρα από αυτές τις αλλαγές στο επίπεδο της θάλασσας θα και έχουμε και τα ιστορικά ακραία φαινόμενα λόγω των πολύ εντόνων καταιγίδων. αυτά τα φαινόμενα στο μέλλον θα γίνουν πιο συχνά. Υπάρχει πιθανότητα ορισμένα από αυτά Αντί να συμβαίνουν μια φορά τον αιώνα, να συμβαίνουν μια φορά το χρόνο. Και αυτό θα συμβαίνει στην διάρκεια παλήριας ε, με πολύ έντονες καταιγίδε και πόλεις οι οποίες είναι παράκτης ή τα μικρά νησιωτικά κράτη θα απειλούνται κάθε χρόνο μέχρι το 2050, ειδικά αν δεν υπάρξει ισχυρή προσαρμογή και όπως είπα και στις στα χαμηλότερα υψόμετρα. Έχουμε κάνει κάποιες εκτιμήσεις κινδύνου ε, για διάφορες περιοχές που επηρεάζονται από την ε, άνοδο του επίπεδου της θάλασσας και έχουμε μία σύγκριση στην αριστερή στήλη που δείχνει τις σημερινές προσπάθειες προσαρμογής και την ανάπτυξη του κινδύνου εάν προχωρήσουμε σε φιλόδοξη προσαρμογή και προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τις ακτογραμμές. Υπάρχουν διάφορες ε, παράκτιες πόλεις όπου βλέπουμε πως ο κίνδυνος μπορεί να μείνει στο κίτρινο πεδίο ακόμα και ε, μέχρι το τέλος του αιώνα. Γιατί αυτό είναι ο χρονικός ορίζοντας στον οποίο έγινε αυτή η μελέτη. Εάν πάμε όμως σε μεγάλα τροπικά γεωργικά δέλτα, θα δούμε ότι μειώνεται η επιτυχία. Και τα πράσινα εκείνα κομμάτια δείχνουν πόσο η προσαρμογή μπορεί να γίνει, αλλά και πόσο μπορεί να, και να επιβληθεί η μετεγκατάσταση από τη στιγμή που μακροπρόθεσμα δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν ε, τα συγκεκριμένα μέρη. Υπάρχουν πολλές κοινωνικές προκλήσεις. Οι άνθρωποι οι οποίοι εκτίθενται περισσότερο και είναι πιο ευάλωτοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν θα πρέπει να σκεφτούμε τους χρονικούς ορίζοντες ε, για αμετάκλητες αλλαγές σε αυτά τα συστήματα. Είναι μακρύτεροι οι ορίζοντες από ότι οι κυβερνητικές ρυθμίσεις. Δεν υπάρχει δηλαδή αντιστοιχία Οι κυβερνητικές ρυθμίσεις είναι, είναι πολύ κατακαιρματισμένες και δεν δίνουν ολοκληρωμένες απαντήσεις σε αυτούς τους αυξανόμενους ε, κινδύνους οι οποίοι ε, εξελίσσονται αλυσίδωτα. Οι δυνατότητες ανταπόκρισης των κυβερνητικών συστημάτων δεν είναι αρκετά συντονισμένοι, ούτε αρκετά γρήγοροι, ούτε αρκετά στεναροί. Για να συνοψίσουμε αυτή την έκθεση, για το 80% ε, της επιφάνειας της γης, οι κλιματικές αλλαγές επηρεάζουν ε, τα συστήματα συντήρησης της ζωής από τις κορυφές των βουνών μέχρι τα βάθη των ωκεανών και το βλέπουμε αυτό από την τήξη των πάγων στα ψηλά βουνά η τήξη του πάγων ε, των, των παγετώνων της Αρκτικής και της Ανταρκτικής, το λιώσιμο των ε, θαλάσσιων πάγων, βλέπουμε τα θαλάσσια κύματα, θερμά κύματα και μετά βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό για την απώλεια οξυγόνου στους ωκεανούς. Αυτές οι αλλαγές θα συνεχιστούν για τις επόμενες γενναίες ανάλογα με τις αποφάσεις που θα λάβουμε τώρα και ε, για να δούμε μια γενική εικόνα σε με αυτές τις τρεις ειδικέ εκθέσεις που ενέκρινε το IPCC το τελευταίο χρόνο είναι μια ανευπροηγουμένου προσπάθεια ώστε να ενημερωθεί η κοινωνία, να μειωθεί ο αντίκτυπος, οι κοινωνικές επιπτώσεις κάθε χρόνος μετρά, κάθε επιλογή μετρά και ακόμη πιο σημαντικό είναι η πολιτική και η κοινωνική βούληση έχουν σημασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Um, Ευχαριστούμε. Ο κατάλογος για το ΚΑΤΣΤΙΑΙ είναι ανοιχτός. Ε, έξι, εφτά οι ομιλητές. So, um... E Ξεκινάμε με το ΕΛΚ. Πίτερ Φαντάλε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ για την τόσο σημαντική αυτή έκθεση που μας παρουσιάσετε, την περίληψη της. Εγώ είμαι στην Επιτροπή Αλίας και γι' αυτό και με ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα όσα λέτε, όπως επίσης και τα θέματα της υπεραλίευσης. Αν κατάλαβα καλά λοιπόν, βλέπω ότι σε ολόκληρη τη γη, σε όλες τις θάλασσες, ε, στις νότιες, ε, στις βόρειες, παντού, αλλιεύονται λιγότερα ψάρια, κατά 50% ουσιαστικά, σε σχέση με το 1900 ας πούμε. Οπότε η ερώτησή μου είναι, καλά τα έχω καταλάβει και αν είναι έτσι, τι σημαίνει αυτό για τον ηλευτικό τομέα στη Βόρεια Θάλασσα, για παράδειγμα, αλλά και τι σημαίνει και για τις επιπτώσεις επί του κλίματος. Εφόσον οι εκπομπές ε, αερίων του θερμοκηπίου αυξηθούν, θα μπορούμε να αλλιεύουμε ακόμα. Θα υπάρχουν ακόμα ψάρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ντάλη. Πρέπει να παρέμβω γιατί διάβασα την έκθεση και σοκαρίστηκα με αυτά που άκουσα. Για μένα κυρίως που έρχομαι από, είμαι από ένα νησί. Έχουμε παράκτιες πόλεις και Ακούμε τώρα δηλώσει που λένε ότι συνεχίζεται να αυξάνεται η στάθμη της θάλασσας και ότι θα έχουμε πολύ ψηλά επίπεδα της επιφάνεια τη θάλασσας όταν θα αρχίσουν αυτά τα έκτακτα φαινόμενα. Ε, αυτά είναι ε, πράγματα που όταν ε, τα ακούει κάποιο που είναι από νησί μπορεί να θεωρεί ότι εκεί που θα γινόταν κάτι σε 100 χρόνια το βλέπει να γίνεται τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω κυρίως για τα ευρήματα, γιατί πιστεύω ότι και οι ωκεανοί έχουν πολύ μεγάλο δυναμικό, κυρίως στη φορά τις δράσεις με βάση τους ωκεανούς. Οι κλιματικές δράσεις με βάση τους ωκεανούς μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση κατά 21% που μπορεί να επιτευχθεί όταν μιλούμε για τις γενικές μειώσεις των εκπομπών. Και ταυτόχρονα έχουμε και θέματα με, την, ε, ε, με τη χρήση του άνθρακα για τις ε, θαλάσσιες μεταφορές και τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Βεβαίω εδώ χρειάζεται περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερε επενδύσει. Όλα αυτά λοιπόν συνδέονται, σχετίζονται με του ωκεανού και θα ήθελα να μα πείτε την γενική σα άποψη. Πέραν των ευρημάτων τη εκθέσεω για το πώ βλέπετε δηλαδή τα πράγματα να εξελίσσονται, και πώς βλέπετε να εξελίσσεται η τεχνολογία. Αν δηλαδή υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει πιθανότητα να γίνει πιο γρήγορα αυτή η αύξηση της στάθμης των ωκεανών σε σχέση με το πόσο, πότε θα γινόταν πριν από λίγα χρόνια. Ευχαριστούμε. Συγγνώμη. Ναι. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και χαίρομαι γιατί το 2014 μαζί με άλλα μέλη της κοινωνίας των πολιτών, φτιάξαμε την πλατφόρμα Επιστήμη και Κλίμα. Τότε δεν μιλούσαμε για τους ωκεανούς όταν μιλούσαμε για την κλιματική αλλαγή και εμείς με μεγάλη περηφάνεια ε, στην COP25 ε, στο Παρίσι καταφέραμε να εισάγουμε και τον όρο ωκεανή στο προήμιο της Συμφωνίας ε, του Παρισιού. Και σωστά, γιατί οι ωκεανοί παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ισορροπία του κλίματος. Ε, δεν είχατε σίγουρα χρόνο να το παρουσιάσετε εδώ, αλλά στην έκθεσή σας το λέτε ότι και οι ωκεανοί αποτελούν μέρος της λύσης. Είναι ένα κεφάλαιο που αφιερώνεται και σε αυτό και νομίζω ότι μπορούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας που οι επιστήμονες συμμετέχουν στη συζήτηση της κοινωνίας των πολιτών αναφερόμενοι σε λύσεις. Θα ήθελα λοιπόν να μας μιλήσετε περισσότερο για τις λύσεις και να αναφερθώ και σε ένα έγγραφο το οποίο δημοσιεύθηκε από μια οργάνωση Ocean for Climate λέγεται το έγγραφο αυτό και εξηγεί πώς και οι ωκεανοί μπορούν να βοηθήσουν για τη λύση. Θα ήθελα να σταθείτε λίγο σε αυτό, γιατί εγώ δυσκολεύομαι να καταλάβω. Όταν σας ακούμε, και όταν βλέπουμε τις καμπύλες των επιστημόνων, καταλαβαίνουμε ότι η δράση μας πρέπει να είναι αμέσως. Όμως, οι ωκεανοί έχουν κάποια αδράνεια. Ακόμα δηλαδή και αν σήμερα αναλάβουμε κάποια δράση, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι ο αντίκτυπος θα είναι ορατός αμέσως, ας πούμε όσον αφορά ε, την αύξηση της στάθμης των υδάτων. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μας διαφωτίσετε για αυτά, για τις λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν για την προστασία των θαλωσίων ε, οικοσυστημάτων, αλλά επίσης να καταλάβουμε λίγο καλύτερα αν δράσουμε κάπως σήμερα αυτό, πότε θα έχει αντίκτυπο στους ωκεανούς. πράσινη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πραγματικά πολύ ανησυχητικό να ακούμε τα αποτελέσματα αυτά της έκθεσης. Πραγματικά μας ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι και μας ανησυχεί πάρα πολύ το να βλέπουμε τέτοια δεδομένα. Δεδομένου του ότι οι ωκεανοί καλύπτουν το 70%, πάνω από το 70%, της επιφάνειας του πλανήτη και 97% του, των υδάτων του πλανήτη, καμιά φορά αναρωτιέμαι μήπως ε, θα έπρεπε, έπρεπε τον πλανήτη να τον λέμε γη ή να τον λέμε ωκεανό, γιατί ο ωκεανός θα είναι τελικά αυτός που θα συμβάλλει στην προσπάθειά μας να μετριάσουμε και να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή. Αν το κάνουμε εγκαίρως, αν δράσουμε επιγόντως και άμεσα, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μια ε, ισχυρή συνθήκη για τους ε, ωκεανούς που δημιουργούσε ε, περισσότερα δίκτυα για τους ωκεανούς και έβαζε ένα 30% των ωκεανών εκτός ορίων για ανθρώπινες δραστηριότητε. Θα μπορούσε να βοηθήσει κάτι τέτοιο. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μείωνε τουλάχιστον 65% μέχρι το 2030 τις εκπομπές αερίων. Θεωρείτε ότι τέτοια δράση θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Και επίσης, Πρόεδρε, σήμερα το πρωί ήμουν σε μια συνάντηση όπου η αυτή η, η, λίστα των κοινών συμφερόντων περιλαμβάνει α, project όπως εισαγωγή ε, αερίου από την Πενσιλβάνια, από τις ΗΠΑ, όπως είπατε και εσείς, ο κύριος Τραμπ έχει αποφασίσει να απομακρυνθεί από τις κλιματικές συμφωνίες και η Ένωση υποστηρίζει μια χώρα όπως η Ιρλανδία που έχει σκοπό να εισάγει ε, το αέριο της Πενσιλβάνια σε περιοχές στην ε, νότιο-δυτική Ιρλανδία. Όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να πάψουν γιατί πρέπει να κινηθούμε προς τις ε, ανανεώσιμες πηγές. Ευχαριστώ. Ο Κρις Ντέιβις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ω πρόεδρο τη ε, Επιτροπή Αλία, θέλω να δω κάτι καλό από όλη αυτή την συζήτηση. Βεβαίω πρέπει να λάβουμε μέτρα, βεβαίω πρέπει να σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή. Ό,τι και να κάνουμε, ακούμε ότι θα μειωθούν τα αλληλευτικά αποθέματα ε, σε όλο τον ε, πλανήτη. Αλλά ω αποτέλεσμα των δικών μα δράσεων, μέσω υπεραλίευσης κτλ. Τα αποθέματα έχουν μειωθεί δραματικά τα τελευταίο, τον τελευταίο αιώνα. Καμιά φορά έχουμε δει μείωση του 80% ή και μεγαλύτερη. Υπάρχει λοιπόν οποιοδήποτε λόγος αν πάρουμε τα μέτρα και σταματήσουμε την υπεραλίευση και αφήσουμε τα, να αναζωογονηθούν τα αποθέματα να καταλήξουμε σε περισσότερα αποθέματα. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ακόμη και ότι, ό,τι και να κάνουμε τώρα να καταλήξουμε σε περισσότερα αποθέματα λευτικά από ό,τι έχουμε τώρα, παρά την κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ. Μάικλ Μπλος για τους πρασίνους και πάλι. Ευχαριστώ. Είναι τρομακτικά αυτά που βλέπουμε στην έκθεση και ευχαριστώ που καλέσατε πρόεδρε τους ε, ε, εμπειρογνώμονες για την παρουσίαση αυτή. Είπαμε ότι ε, ένα μέτρο θα αυξηθεί η στάθμη της θάλασσας ε, μέχρι το τέλος του αιώνα, πέντε μέτρα ίσως μέχρι το 2300. Για το οικονομικό κόστος μπορείτε να μας πείτε κάτι και επίσης μήπως μπορείτε να μας πείτε για το κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πόσο θα είναι ο αντίκτυπος και ποιο είναι το κόστος των ε, άμεσων επικουσών δράσεων για να αποφύγουμε αυτά τα φαινόμενα. Η επένδυση δηλαδή πόση θα είναι. Και επίσης, μήπως μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσοι άνθρωποι θα επηρεαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτή την αύξηση ενό μέτρου τη στάθμη τη θάλασσα και σε ποια κράτη-μέλη. Um, um, θα θέλαμε όλε αυτέ τι ε, λεπτομέρειες να μας τις πείτε για να ξέρουμε όσο δυνατόν περισσότερα στοιχεία για το πότε θα μα ε, μας χτυπήσουν όλα αυτά τα φαινόμενα. Renew, Pierre Renew, Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Δεν θα επανέλθω σε όσα είπαν οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Αλίας, αλλά Κάτι ακόμα. Θα υπάρχουν περισσότερα, λιγότερα ψάρια, αυτά ρώτησε ο Κρις Ντέβης. Το αν θα υπάρχουν περισσότερα, λιγότερα, ε, τι σημαίνει. Εμείς καταλαβαίνουμε από αυτά που λέτε, είναι ότι θα αλλάξει η κατάσταση. Θα υπάρξει αλλαγή, όχι μόνο ποσοτική, αλλά και ποιοτική. Δηλαδή, τα είδη, τα ίδια θα αλλάξουν. Το λένε και ήδη οι αλείς, ότι υπάρχει η αλλαγή με την έννοια ότι τα αποθέματα κυκλοφορούν και φεύγουν από ένα μέρος και πηγαίνουν σε κάποιο άλλο και τα βρίσκουμε αλλού, μετακίνονται πόσο, 5 χιλιόμετρα, 40 χιλιόμετρα σύμφωνα με κάποιες ε, έρευνες πηγαίνουν πιο βόρεια. Οπότε θα πρέπει σε αυτή τη θητεία να αποφασίσουμε για την κοινή αλλιευτική πολιτική. Προς το παρόν Αυτά που εμφανίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια αξιολόγηση, αντί και μια προσαρμογή. Εγώ θα έλεγα ότι η κοινή μας ελευτική πολιτική θα είναι μέχρι το 2030, οπότε εμεί πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί το 2040 φαίνεται ότι η ίδια η δομή των διατροφικών αλυσίδων που περιλαμβάνουν ε, ε, ψάρια ε, θα έχουν αλλάξει. Γιατί τα ίδια τα λιεύματα θα έχουν αλλάξει. Οπότε δεν πρέπει μόνο να κάνουμε μια αξιολόγηση, αλλά να δούμε σε βάθος την κατάσταση, ώστε να προσαρμοστεί ένας κλάδος, ο οποίος, κοιτάξτε, σήμερα Πόσο κρατά ένα σκάφο, 30, 40 χρόνια. Σε 40 χρόνια όμω θα ψαρεύει ω κάτι εντελώ διαφορετικό από αυτό που ψαρεύει σήμερα. Ευχαριστούμε. Οι δύο τελευταίοι ε, από τους πράσινους, τα πάλους πρώτα. Ευχαριστώ για την έκθεση αυτή. Πολλοί συνάδελφοι έκαναν σχόλια. Είναι τρομακτικά αυτά που μας λέτε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι που μπορεί να τρομάξει την κατάσταση ακόμα περισσότερο, γιατί για την πέρμαφορο στο, τους αιώνιους πάγους, οι οποίοι ε, λιώνουν όλο και πιο γρήγορα και υπάρχουν κομμάτια που δεν έχουν πια πάγο καθόλου και είμαστε στο Νοέμβριο. Οι εκτιμήσεις ε, αυτές βέβαια εξακολουθούν να είναι θα έλεγα αισιόδοξε γιατί έτσι όπως έχει μειωθεί ο πάγος, υπάρχει περίπτωση να ξαναπαγώσει μέσα στο χειμώνα τόσο πολύ όσο συνέβαινε παλιότερα. Αυτό μπορούμε να το δούμε με δορυφόρους. Και όσον αφορά την ε, οκενολογική έρευνα, ε, μία ερευνήτρια είχε πει ότι η Αρκτική σε 750 ppm αρχίζει να ξαναφτιάχνει ε, πάγο, ενώ πριν αυτό γινόταν ήταν στα 315 ppm. Οπότε φοβάμαι ότι η Αρκτική, ρωτάω δηλαδή, με τους ρυθμούς που έχουμε σήμερα και τις θερμοκρατίες που έχουμε σήμερα, Μήπως τελικά είναι αναπόφευτο να εξαφανιστεί ο πάγος εκεί. Χόλγρον Πράσινη. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να συνεχίσω μετά την προηγούμενη ακριβώς ερώτηση. Συνήθως συζητάμε για ένα, ενάμιση, δύο βαθμούς θερμοκρασία, αλλά υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες που λένε ότι ίσως θα έπρεπε να συζητήσουμε περισσότερο για το ποσό του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Ο James Falkton πριν από μερικά χρόνια είχε πει ότι το όριο είναι 350 ppm διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και δεν πρέπει να ξεπεραστεί αυτό. Και αυτό είναι και το όριο που και το Ινστιτούτο της Στοκχόλμης αναφέρει επίσης. Θα συμφωνούσατε λοιπόν ότι θα έπρεπε να είμαστε στα 350 στα τέλη του αιώνα αυτού προκειμένου να μπορέσουμε να κρατήσουμε την θέρμαση του πλανήτη σε τέτοια επίπεδα που να μπορούμε να τη χειριστούμε. Ενώ τώρα είμαστε στα 410 ppm και έχουμε αύξηση 3 ppm το χρόνο. Οπότε καταλαβαίνετε που θα φτάσουμε σε λίγα χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ωραία. Δέκα λεπτά λοιπόν έχετε εσείς στη διάθεσή σας για να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Θα προσπαθήσω και θα αρχίσω με την Αλία. Σίγουρα με τις αλλαγές που διαπιστώνουμε, ναι, μπορώ να απαντήσω, θα έχουμε λιγότερα ψάρια στο μέλλον. Και ανάλογα με το βαθμό της κλιματικής αλλαγής και το μέσο όρο της αλλαγής, αυτές οι αλλαγές θα είναι μεγαλύτερες ή λιγότερες. <coughs> Αυτή είναι η συζήτηση. Και στη συζήτηση με τη γη είδαμε ότι τα ίδια και για την βιοπικιλότητα. Τα ίδια ισχύουν λοιπόν και για τους ωκεανούς. Υπάρχουν συναντήσεις κάθε χρόνο. Πριν από δύο εβδομάδες ήμουν σε μια διάσκεψη για τους ωκεανούς που φιλοδοξεί να απομονώσει προστατευμένες περιοχές για να προστατεύσει εκεί τους φυσικούς πόρους. Προκειμένου οι θαλάσσιοι πόροι να μπορούν να μετακινούνται και να εξακολουθούν να είναι προστατευμένοι. Ένα μεγάλο μέρος των ωκεανών πρέπει να προστατευτεί με αυτόν τον τρόπο. Φτάνουμε στο 10% που είναι ο στόχος μας για τις εθνικές προσπάθειες και αυτό σίγουρα θα βοηθήσει. Όμως αυτό που πρέπει συγχρόνως να πούμε και ισχύει για κάθε προσπάθεια αποκατάστασης ε, κορολιογενών ε, περιοχών είναι ότι οι προσπάθειες αυτές μπορεί να είναι μάταιες αν δεν πετύχουμε να περιορίσουμε τη θέρμανση του πλανήτη. να μην υπάρξει αύξηση της θερμοκρασίας λοιπόν, πέρα από το 1,5 βαθμό, γιατί αυτό είναι προϋπόθεση προκειμένου να πετύχουν αυτά τα διάφορα μέτρα προστασίας στο θαλάσσιο χώρο. Ήδη πρόκειται για ένα μεγάλο κομμάτι των κορελογενειών ε, περιοχών. Πρόκειται για την ε, μετακίνηση της ε, θαλάσσιας ζωής που εξαρτάται από τις θερμοκρασίες και αυτό έχει να κάνει και με αλλαγές στην Αρκτική. Οι πάγοι στη θάλασσα θέλουμε να παραμείνουν και το καλοκαίρι, αλλά δεν θα παραμείνουν αν συνεχιστεί η θέρμαση του πλανήτη. Και δεν μας ε, εκπλήσει που η πολιτική συζήτηση επικεντρώνεται ε, σε αυτό το όριο της θερμοκρασίας, τον 1,5 βαθμό. Τώρα έτσι απαντάω, νομίζω, στις ερωτήσεις σας για την αλία. Έτσι κι αλλιώς ένα είναι το συμπέρασμα, συνολικά. Ότι πρέπει να υπάρξει σταθεροποίηση του κλίματος αν θέλουμε να προστατεύσουμε ε, τους σπόρους. Ρωτήσατε και τα μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αναφέρονται στην έκθεσή μας για τον ανάμεση βαθμό, όπου μιλάνε για τη μείωση των εκπομπών το 2020 και το 2030 σε σχέση με το 2010 και το 2050 να έχουμε ουδετερότητα όσον αφορά το αποτύπωμα άνθρακα. Οπότε, ναι, υπάρχουν διαθέσιμα σενάρια, τα οποία μπορούν να κατευθύνουν τις πολιτικές σας φιλοδοξίες. Σε σχέση με τη Συμφωνία του Παρισιού. Υπάρχει η Συμφωνία του Παρισιού και τώρα το θέμα είναι η υλοποίησή της. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Και ναι, υπάρχουν μέρη ακόμα και στην Ευρώπη που απειλούνται. Και εγώ ζω σε μια τέτοια περιοχή που είναι χαμηλά στο επίπεδο της θάλασσας. Δεν μπορώ να σας δώσω νούμερα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το οι άνθρωποι δηλαδή θα επηρεαστούν. Το θέμα είναι πότε θα πετύχουμε την ε, προσαρμογή. Οι ακτές έχουν ακόμα περιθώρια και μπορούμε τα φράγματα να τα μεγαλώσουμε, να τα ψηλώσουμε, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια ακραία φαινόμενα αύξησης του επίπεδου της θάλασσας. Τώρα για το πότε θα συμβεί αυτό και πώς, υπάρχει μεγάλη βεβαιότητα για την αύξηση του επίπεδου της θάλασσας. Οι αριθμοί που δίνουμε είναι οι καλύτερες εκτιμήσεις που διαθέτουμε. Αλλά υπάρχει αβεβαιότητα για διάφορα θέματα, γιατί εξαρτάται κατά πόσο θα επιταχυνθεί ακόμα περισσότερο η άνοδος των υδάτων δεν ξέρουμε αν αυτό θα γίνει με τον 1,5 βαθμό ή με 4. Το θέμα είναι ότι τα νούμερα τα οποία έχουμε τώρα ανταποκρίνονται ε, σε στοιχεία που έχουμε από το παρελθόν. Η ακρίβεια βέβαια εξαρτάται από το τι θα λάβει υπόψη, αν θα λάβει υπόψη όλα τα δεδομένα που υπάρχουν πλανητικά. Υπάρχει το απόθεμα των 65 μέτρων που λέει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει κανείς ακριβείς προβολές. Πρέπει να καταλάβει κανείς όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας που οδηγεί στην τήξη των πάγων. Ναι, μπορούν οι ωκεανοί φυσικά να συνεισφέρουν στο μετριασμό και στην έκθεση αυτή έχουμε εξετάσει λύσεις που βασίζονται στη φύση. Αλλά τα νούμερα για τις παράκτιες περιοχές και διάφορα οικοσυστήματα που μπορούν να αποκατασταθούν δεν έχουν πάνω από 0,5% το χρόνο. Οπότε όταν μιλάμε για μείωση, αυτή πρέπει να γίνει. Γιατί αν δεν γίνει, τότε οποιαδήποτε προσπάθεια είναι μάτι. Η αποθήκευση του άνθρακα στους ωκεανούς είναι κάτι που δεν έχουμε ακόμα εξετάσει αρκετά. Αλλά υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Που δεν έχουν όμως αξιολογηθεί οριστικά ακόμα. Αλλά θα το κάνουμε αυτό με τους αδέρφους από τις ομάδες εργασίας. Τώρα για το πάνω από 20% συνεισφορά στη εναλλακτική ενέργεια δηλαδή από τους ωκεανούς με την εκμετάλλευση του ανέμου, σύμφωνα με το IPCC, πάλι θα γίνει σχετική αξιολόγηση στην ομάδα εργασίας 3. Οι εκπομπές από την αυτιλία. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Όπως και από την ε, αεροπορία. Και εγώ είμαι από μια χώρα όπου γίνεται ευρεία συζήτηση για τη δυνατότητα χρήση συνθετικών καυσίμων, συνθετικού ντίζελ ή υδρογόνου ή ακόμα παραγωγής υδρογόνου από φυσικό αέριο και αποθήκευση του άνθρακα. Είναι πράγματα που συζητιούνται. Είναι εναλλακτικές επιλογές που δεν έχουν εξεταστεί επαρκώς ακόμα και δεν έχουν οριμάσει τεχνολογικά. Αν όμως θέλεις φιλόδοξη μείωση, υπάρχει η ελπίδα να πετύχουν αυτά. Αν θα πετύχουν τώρα ε, τόσο γρήγορα όσο χρειάζεται για να πετύχουμε τους στόχους του Παρισιού, αυτό εξαρτάται από την πολιτική βούληση και την βούληση της κοινωνίας. Υπάρχουν επιλογές που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και να εκμεταλλευτούν. Στην ειδική μας έκθεση για τις λύσεις έχουμε εξετάσει λύσεις από τη φύση. Και έχουμε και λύση για την προστασία των ακτών. Υπάρχει ένας πίνακας για τους πολιτικούς που αναφέρει διάφορες αναλυτικές λύσεις για την προστασία των ακτών. Τέλος, Όσον αφορά τη συγκέντρωση του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, ναι, γνωρίζω ότι συζητήσει αυτές. Κάποιοι μιλάνε ναι, για την Αρκτική και για τα 350 ppm, αλλά τότε πρέπει να έχουμε τεχνολογικές εξελίξεις επιτυχής που να αξίζει τον κόπο να τις εκμεταλλευτούμε ώστε να μεταφερθεί από την ατμόσφαιρα το διοξείδιο του άνθρακα, αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί. Αυτά έχω να πω προς το παρόν. Uh, Ευχαριστώ. Ένα τελευταίο χειροκρότημα για όλους σας. Thank you very much uh, again for the message and for your work. I suggest uh, a two minutes break so that we can have the να κάνουμε ένα δίλεπτο διαλυματάκι για να φύγουν όσοι πρέπει, να μείνουν όσοι πρέπει και να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Dear colleagues, I will ask you to get back to your seats. Λοιπόν, συνάδελφοι, καθίστε, παρακαλώ. Να ξεκινήσουμε και να περάσω κι εγώ στα γαλλικά. Μη λες όχι, μη λες όχι. Pourquoi, pourquoi Donc nous votons Commençons par le vote sur la question orale au Conseil. Λοιπόν, πάμε να ψηφίσουμε για την προφορική ερώτηση του Συμβουλίου για την COP15. Προφορική ερώτηση λοιπόν για την COP15, για τη βιοπικιλότητα. Άρχεται την ψηφοφορία. It's Δεν δουλεύουν τα συστήματά μας. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η προφορική ερώτηση. Πάμε στην προφορική ερώτηση για το Ευρωπαϊκό Έτος για τις πιο πράσινες πόλεις 2021. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περάμε στην προφορική ερώτηση για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Πέρας, από ε, την ψηφοφορία. Le vote est clos. Πέρας ψηφοφορίας. Adopté. Εγκρίνεται. Son, euh, au vote sur... les... Περνάμε στο παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιά. Άρχεται η ψηφοφορία. Le vote est clos. Πέρας ψηφοφορίας. Très bien. Nous passons maintenant au Εγκρίνεται. Πάμε στο ψήφισμα για την COP25. Δεν θα γίνει στη Χιλή πλέον, αλλά στην Ισπανία. Θα γίνουν εκεί οι βασικές ε, απαραίτητες τροποποιήσεις. Το κείμενο θα τροποποιηθεί. Η Προεδρία θα είναι χιλιανή, αλλά η διάσκεψη θα γίνει στη Μαδρίτη. Πάμε στην ψηφοφορία. Παράγραφος 1, τροπολογία 13. Α, είναι προφορική. Είναι προφορική. C'est bon So, paragraph 1. Παράγραφος 1. Προτροπολογία 35. Ποιος είναι υπέρ? Υπέρ. Υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Απορρίπτεται. Ποιος απέχει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Συνάδελφε, ευχαριστώ. Η προσθέμενη αξία σας απεδείχθη. Λοιπόν, τροπολογία 36, παράγραφος 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. So it's not working? No, but that's okay. It's not best. Εγκρίνεται. Τροπολογία Παράγραφος 1, τροπολογία 37. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην παράγραφο 2α, τροπολογία 45. Ποιος είναι υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Α, να το ελέγξουμε. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. No, sorry. <laughs> Πέρας ψηφοφορίας. Τροπολογία 46 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 48 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρα Πέρας ψηφοφορίας. Έγκρινεται. Χωρίς την ψηφοφορία για την τροπολογία 50. Για το πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται. Ποιος είναι υπέρ του δεύτερου τμήματος. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 54. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 55, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, αλλά να το ελέγξουμε κιόλας. Πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Συμβιβαστική πρόταση 14, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 4, τροπολογία 57. 57, 57 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 5. Τροπολογία 62. Υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται η τροπολογία. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 75. Υπέρ. Κατά. Ποιος είναι υπέρ και ποιος είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. 79. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 84, υπέρ, κατά. Ε, δεν είναι σαφές από τους οριστές. 84, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 85. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η τροπολογία. 87. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 88. Υπέρ κατά. Ηλεκτρονικά παρακαλώ να ψηφίσουμε την 88. Le vote Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 102. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλα, έχουμε και πάλι ηλεκτρονικά. Την 102 ψηφίζουμε. So the vote is closed. ο ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 105. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Την 103 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Body's closed. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 106. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 108. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Την 108. Okay. Sorry. It's clear. Adopted. Εγκρίνεται. 109. Χωριστή ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Ποιο είναι υπέρ. Ποιο είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεν κατάλαβα οι σοσιαλιστές τι ψήφισαν, υπέρ, άρα εγκρίνεται μάλλον. Εντάξει, μπορείτε και να αλλάξετε γνώμη, ε. Λοιπόν, ελέγχουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα της 109. Εγκρίνεται. 110. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική πρόταση 15. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 118. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 118. Rejeté. Απορρίπτεται. Τροπολογία 119. Υπέρ. Ποιος είναι κατά. Ποιος απέχει. Απορρίπτεται. 120. Υπέρ κατά, αποχές, να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά, νομίζω απορρίπτεται ωστόσο. Rejected. Όντως απορρίπτεται. 121. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 124. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Sorry. Λάθος, λάθος. Καταπίπτει. Καταπίπτει αν έχει εγκριθεί 123 και έχει εγκριθεί 123, οπότε 124 καταπίπτει. Πάμε στην 125. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 128 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 129 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 130 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 131 υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. 132. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 133. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 134. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται, εγκρίνεται. 140 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 141 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 147. 147 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 148 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. εκατόν πενήντα, ε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 151 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 153. Χωριστή ψηφοφορία, πρώτο μέρος, ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά, να το ελέγξουμε, νομίζω απορρίπτεται. Rejected. Απορρίπτεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Την 155 ψηφίζουμε. Πέρα closed. Πέρας ψηφοφορίας Απορρίπτεται. Τροπολογία 156. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 158. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 157. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. 157. Την 157. Α, όχι. Καταπίπτει. Άρα που πάμε. Στην 159. Συγγνώμη, συγγνώμη. Πάμε στην 159. Η 157 καταπίπτει. Υπέρ για την 159. Κατά. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 159 αυτή τη φορά. closed. Πέρας Εγκρίνεται. Συμβιβαστική πρόταση παριθμών 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκατόν εξήντα ένα. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. What is closed. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 170. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 171 υπέρ. 171 είπα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 171 λοιπόν. Hmm. Sorry about that. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Συμβιβαστική πρόταση 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 182. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρα is closed. εγκρίνεται η τροπολογία 182. Προφορική τροπολογία 183. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να το ελέγξουμε. Αν θέλετε, το ελέγχουμε. Εντάξει, απορρίπτεται. Εκατόν ογδόντα έξι. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 187. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 188. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 194. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 195. Υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. 196 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 199 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 200 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Πέρα. closed. Πέρας. Απορρίπτεται. Διακόσια ένα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε και πάλι ηλεκτρονικά. Τη 201. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 203. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Celui-là aussi tombe 205. C'est ça. Amendement 205. 205. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 206. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 208. Υπέρ. Λοιπόν, από την αρχή, 208, υπέρ, κατά, να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται. Ξεκάθαρα απορρίπτεται. <laughs> Amendement 209. Τροπολογία 209. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε να ψηφίσουμε την 214 γιατί δεν έχει εγκριθεί η συμβαστική 16. 214. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2-10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 213. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 215. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 211 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 212 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 228. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Συμβαστική 11 πρώτα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 228 τώρα λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 235 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13α υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την συμβαστική 13α. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 244. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 245 καταπίπτει γιατί 153 έχει εγγραφεί. Πάμε στην 246. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.48 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται νομίζω, αλλά να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Le 247, Απορρίπτεται. 252. 252. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το EPP είναι υπέρ. Λοιπόν, ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 252. Rejected. Απορρίπτεται. 254 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 253 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 256 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 257 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.55 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.58 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.59 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.60 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Έγκρινεται. 2.61 υπέρ. Κατά. Πάλι ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. Δεν δουλεύει το... η συσκευή σας. Συν ένα λοιπόν. Συν ένα κατά. Εντάξει. 2,62. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2,63 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 264 υπέρ, κατά, αποχές έγκρινεται. 265 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 266 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 267 υπέρ, κατά, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται. 2.44 υπέρ. Όχι. Συγγνώμη, συγγνώμη, δεν έχω χρώματα εγώ στο δικό μου το αντίτυπο. Πάμε στη 2.68 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2,69 υπέρ. Κατά. Ε, αποχές εγκρίνεται. 2,70 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2,71 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2,72 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Έγκρινεται. 276 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 274 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. 274. Τη 274. It's Απορρίπτεται. Ε, ψηλά τα χέρια σας, να σας βλέπω. 2,77 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2,78 υπέρ, κατά, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Adoptez. Εγκρίνεται. 2. 79. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.80. Υπέρ. 2.81. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 283 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 284 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 285 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 286 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 287 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε μπλοκ για τις ε, τροπολογίες ήτρε. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Επίσης το ίδιο για τις τροπολογίες ΔΕΒΕ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. ΔΕΒΕ 1 έως 3, 5 7 και 12 15. Ψηφίζουμε τώρα. Δεν ψηφίζουμε μάλλον τις επόμενες. Και πάμε στις ε, ε, αιτιολογικές σκέψεις. 12. Όχι τη 12. Πάμε στην 7. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 16, τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ο 11 υπέρ. Κατά.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 στους ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ορίζεται. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 δεν έχει εγκριθεί, άρα ψηφίζουμε την τροπολογία 22. 22 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Rejeté. Απορρίπτεται. Είκοσι Υπέρ. Κατά. Από... Ελέγχουμε και πάλι ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Okay. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Secret You can blame the secretariat. Η γραμματεία, η γραμματεία αυτή. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία και πάλι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το ψήφισμα. Συνεχίζουμε. Περνάμε στις αντιρρήσεις. Αντίρρηση για το βαμβάκι. LL25. Ε, ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίθηκε η αντίρρηση. Τώρα, αντίρρηση για την γενετικά τροποποιημένη σόγια ΜΟΝ 89788. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Τώρα, αντίρρηση για διάφορα αραβόσιτα γενετικά τροποποιημένα. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε η αντίρρηση. Τελευταία ψηφοφορία για άλλους γενετικά τροποποιημένους αραβόσιτους, BT11 κλπ. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της φοφορίας. Εγκρίθηκε. Τώρα.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 Dear colleagues, we still have... Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ακόμα ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ξέρω ότι κουραστήκατε και ότι η ώρα περνάει. Λοιπόν, αν θέλετε να αποχωρήσετε, αποχωρήστε γρήγορα και σύχως. Θα συζητήσουμε τώρα την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατικά και εμπορικά οχήματα και πρόσβαση σε πληροφορίε επισκευή και συντήρησης οχημάτων. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα απ' όλα, την Γενική Διεύθυνση GROW και μετά στην εισηγήτρια, την Έστερ Ντελάνγκε. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα. Πέντε λεπτά παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλους και ευχαριστώ που βάλατε αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Να μιλάτε πιο κοντά στο μικρόφωνο, παρακαλώ. Και οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές εδώ στην αίθουσα, μην κάνετε πηγαδάκια εδώ, ησυχία, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Αν θέλετε να αποχωρήσετε, φύγετε. Αλλιώς, σιωπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που δώσατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να παρουσιάσει την ε, πρόταση αυτή του κανονισμού. Θα περάσω στις διαφάνειες που έχουμε ετοιμάσει, επειδή είναι πολύ τεχνικό το θέμα. Θα εξηγήσω τις αιτίε, ποιες είναι οι προθέσεις και γιατί πράγμα συγκεκριμένα μιλάμε με τη συναπόφαση επί του κανονισμού αυτού. Λοιπόν, ο κανονισμός αυτός και είναι σημαντικό να δώσουμε το πλαίσιο στη σημερινή συνάντηση. Στις 10 Μαρτίου 2016 ενέκρινε τον κανονισμό αυτό για τις εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης που ήταν ένας πολύ σημαντικός ε, κανονισμός γιατί μας επέτρεπε να περάσουμε από τις δοκιμές στο εργαστήριο σε δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες. Ο κανονισμός αυτός λοιπόν που εγκρίθηκε το 2016 συμπληρώθηκε από έναν άλλον την επόμενη χρονιά που εισήγαγε αυτό που ονομάζουμε παράγοντες συμμόρφωσης. Οι πολλαπλασιαστές δηλαδή των ορίων που είχαν ε, τεθεί σε άλλες νομοθετικές πράξεις για να λάβουμε υπόψη μας τεχνικές και στατιστικές αβεβαιότητες που αφορούν τη διαφορά των δοκιμών σε εργαστήριο με τις δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες. Αυτά ήταν τον Απρίλιο του 2016. Στον κανονισμό αυτό, σχετικά με τους παράγοντες συμμόρφωσης και όχι με τις πραγματικές δοκιμές αυτές, ε, κάθε αυτές, έγιναν ε, σε διάφορες πόλεις, ε, Παρίσι, Μαδρίτη και Βρυξέλλες, που προσέβαλαν τον κανονισμό και ιδιαίτερα τους παράγοντες συμμόρφωσης λέγοντας ότι δεν είχε την εντολή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το κάνει αυτό. Πήγαμε λοιπόν στο δικαστήριο αυτές οι πόλεις και περιμέναμε την απόφαση του δικαστηρίου για να δούμε τι λέει το κείμενο του δικαστηρίου. Συγχρόνως όμως, η Επιτροπή όμως αποφάσισε να κάνει έφεση στην απόφαση του δικαστηρίου. Αυτή είναι η κατάσταση πραγμάτων. Η, την Επιτροπή της στήριξε η Γερμανία και η Ουγγαρία και το Γενικό Δικαστήριο είπε ότι σε ένα χρόνο θα κατέληγε στην ε, απόφαση, αλλά επειδή υπάρχει η έφεση, η διαδικασία κρατάει περισσότερο. Σήμερα γνωρίζουμε ότι το δικαστήριο δεν πρόκειται να αποφασίσει για την ε, έφεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από το δεύτερο εξάμεινο του 2020. Οπότε, και εδώ έρχομαι στο σχέδιο κανονισμού που συζητάτε σήμερα, προκειμένου να διασφαλιστεί βεβαιότητα νομική για τους διάφορους παίκτες και για να ακολουθήσουμε και αυτά που είπε στην πρώτη του απόφαση το δικαστήριο, ε, υπάρχει πρόταση από την Επιτροπή για το κείμενο που έχετε μπροστά σα. Και αλλάζει δηλαδή ο κανονισμός 715 του 2007 που βάζει όρια για τα οξύδια του αζότου, για τα σωματίδια, το οξύδιο του άνθρακα και συνολικά για όλα αυτά και τους υδραγωνάθρακες. Και έτσι εμείς περιορίζουμε τους παράγοντες συμμόρφωσης, αυτοί δηλαδή που είχαν κάποια στατιστική αβεβαιότητα και εκείνα που είχαν να κάνουν με τεχνικές αβεβαιότητες, τα βάζουμε στην συναπόφαση, γιατί είπε το δικαστήριο ότι η Επιτροπή δεν είχε την αρμοδιότητα να το κάνει ή γιατί οι παράγοντες ε, συμμόρφωσης είναι πολλαπλασιαστές, πρέπει, είπε, να υπάρχει συναπόφαση. Αυτό είναι λοιπόν το κύριο θέμα για τη συναπόφαση. Εδώ είναι οι παράγοντες συμμόρφωσης που σας έλεγα, που αντικατοπτρίζουν τις τιμές που αρχικά είχαν προταθεί. Εμείς προτείνουμε ένα περιθώριο για τις τεχνικές αβεβαιότητες που είναι ε, χαμηλότερο από τα αρχικά γιατί ξέρουμε ότι το περιθώριο αυτό είναι χαμηλότερο από το 1,5, γι' αυτό έχουμε τις τιμές 1,43 και συνεχίζεται το έργο ακόμα και σήμερα. Η Επιτροπή είπε ότι η αναθεώρηση των τεχνικών περιθωρίων θα γίνεται καθημερινά. Το Κέντρο Κοινό Ερευνών έχει επίσης ε, ξεκινήσει το έργο του και έχουμε ήδη κάποια ε, πρώτα αποτελέσματα, ότι δηλαδή μπορεί να πέσει ακόμα περισσότερο το περιθώριο. Αυτό το ξέρουμε σήμερα, δεν το ξέραμε τον Ιούνιο όταν εγκρίναμε την απόφαση αυτή. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, τα περιθώρια μπορούν να πέσουν ακόμα περισσότερο, στο 0,32. Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα ξέρουμε περισσότερα βέβαια. Τώρα για την πρόοδο στο Συμβούλιο. Βλέπετε ότι οι εργασίες άρχισαν τον Ιούνιο και αυτή τη βδομάδα μάθαμε ότι το Συμβούλιο θα ήθελε να παρουσιάσει πρόταση τέλος Νοεμβρίου στο, στην Κορεπέρ. Οπότε θα μπορέσει στις αρχές επόμενης χρονιάς να ξεκινήσει τριμερής διαλόγου στο Συμβούλιο. Ε, συμπέρασμα. Βλέπετε τα διάφορα άρθρα. Πάντως, το βασικό είναι η αλλαγή που απορρέει από την απόφαση του δικαστηρίου. Δηλαδή, οριοθετούνται οι παράγοντες συμμόρφωσης. Κάτι το οποίο επιτρέπει έγκριση περιθωρίων για τις τεχνικές αβαβαιότητες και τέλος οι υπόλοιπε διατάξεις στο κείμενο είναι διαδικαστικοί κανόνες που χρειάζονται κάποια ενημέρωση βάσει των όσων προβλέπουν οι διαδικασίες κατεξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις. Με δύο λόγια, για αυτούς τους λόγους έχουμε την σημερινή πρόταση. Και από εκεί πέρα είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Η Έστερ Ευχαριστώ πολύ. Η Κομισιόν ξεκίνησε λέγοντας πως πρόκειται για ένα θέμα που είναι εξαιρετικά τεχνικής φύσης και νομική φύσης, αλλά είναι και πολύ ευαίσθητο ζήτημα ε, λόγω όλων των άλλων θεμάτων που συνδέονται με το θέμα αυτό. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μα αν θέλουμε να έχουμε αίσια έκβαση. Θα πω κάποια πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελα εγώ να προσεγγίσω αυτό το ζήτημα. Καταρχάς, θεωρώ πως είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε, γιατί ήδη η λέξη παράγοντας συμμόρφωσης είναι Μόνο και μόνο και να λέμε τέτοια λόγια εδώ είναι αρκού, αρκεί για να αποκαρδιώσει ε, πολλούς. Αλλά ο παράγοντας συμμόρφωσης σημαίνει το να μην υπερβαίνονται τα όρια α, τον, το, το του αζότου και βεβαίως ε, να έχουμε ένα περιθώριο σφάλματος μικρό. Είναι πειρασμός μεγάλος να γίνει αυτή η συζήτηση μόνο για το περιθώριο που σχετίζεται με τον εξοπλισμό δοκιμής αλλά και για το ίδιο το maximum όριο ε, για το οξύδιο του αζότου. Αν κανείς αμφισβητεί στην κατάσταση θα πρέπει αυτό να γίνει για το Euro 7 και όχι σε αυτό εδώ το νομοθέτημα. Θέλω να είμαι σωστή στην προσέγγιση μου, να βασίζομαι στην επιστήμη. Γι' αυτό και η πρώτη μου ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πότε πιστεύετε πως το κοινό ερευνητικό κέντρο, γιατί δεν είμαστε εμείς πολιτικοί, εκείνοι είναι οι πυρογνώμονες, εγώ θα δω τα στοιχεία αλλά για αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να βασιστώ επί των επιστημόνων για να προτείνω με τη σειρά μου μείωση του ορίου. Ε, αλλά η διαδικασία είναι κάπως αόριστη. Θα έχουμε αποτελέσματα τους επόμενους μήνες όπου συζητάμε για αυτό το νομοθέτημα με χαμηλότερο αριθμό. Ποιες είναι οι προσδοκίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το συγκεκριμένο σημείο. Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε αυτό το περίφημο παράγοντα συμμόρφωσης θα πρέπει να είναι σαφής. Να πούμε δηλαδή ότι πρόκειται για ένα όριο το οποίο αφορά τις εκπομπές του ίδιου του αυτοκινήτου, αλλά και ε, το περιθώριο σφάλματος του ε, εξοπλισμού δοκιμής. Και θα πρέπει κάπως να, το να... να είμαστε σαφέστεροι. Αυτό που πρέπει επίση να κάνουμε και νομίζω πως το Κοινοβούλιο θα επιμείνει ότι χρειάζεται μία ε, δυνατότητα αναθεώρησης όταν αυτό χρειάζεται. Δηλαδή, από τη στιγμή που είμαστε έτοιμοι και οποτεδήποτε μπορούμε να κάνουμε αυτό το επόμενο βήμα, να μπορούμε να το κάνουμε και να μην χρειάζεται να δεσμευόμαστε χρονικά. Δεύτερη ερώτηση, γιατί διαφορετικά νομίζω άλλοι θα θέσουν αυτή την ερώτηση, πάλι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ποιο είναι ο χρονικός ορίζοντας για τη συζήτηση για μετά το Euro 6 γιατί θα μιλήσουμε και για τις εκπομπές των ίδιων των αυτοκινήτων, αλλά νομίζω πως αυτό θα πρέπει να γίνει σε αυτό εδώ το νομοθέτημα, αλλά σε νομοθέτημα ξεχωριστό, όπου πρέπει να συζητηθεί αυτό το θέμα. Ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο χρονικός ορίζοντας. Αυτά, Πρόεδρε, και προσβλέπω στα σχόλια όλων όλων, των σκιωδών και τα λοιπά και ελπίζω και από μεμονωμένα ε, συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μίρια Ντελή ε, από τους Σοσιαλιστές, η πρώτη σκιώδης. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και την εισηγήτρια και για Έχουμε επανειλημμένως σε αυτήν την Επιτροπή ε, ακούσει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι δηλαδή τα στάνταρα των εκπομπών θα πρέπει να τηρούνται ε, στον πραγματικό κόσμο και όχι μόνο επί χάρτου. Το 2015 μάλιστα όταν ξέσπασε αυτό το αρνητικό ε, ε, σκάνδαλο του Dieselgate Ήλπιζα πως θα είχαμε έτσι επιταχύνει τις προσπάθειες. Αντί γι' αυτό όμως αντιμετωπίζουμε πάλι τους κατασκευαστές αυτοκινήτων που δεν μπορούν να τα καταφέρουν και δεν μπορούν και να εξοπλίσουν το διζελοκίνητα αυτοκίνητα τα οποία ξεκολουθούν να κυκλοφορούν στους δρόμους μας σήμερα. Και είναι τελείως απαράδεκτο το ότι είχαμε δευτερεογενείς ε, ε, απώλειες που σήμερα περιλαμβάνουν τους παράγοντες ε, ε, συμμόρφωσης ε, που ακόμα συνεχίζουν να εκπέμπουν 168 μικρο χιλιοστόγραμμα. Ε, και, αυτά, και αυτά όλο είναι απαράδεκτο. Ε, αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όπου έχουμε παράγοντα συμμόρφωση, παράγοντες συμμόρφωσης που απλά χρησιμοποιούνται για να, ξαναγραφτεί, να ξαναγραφτούν τα αρχικά όρια περιοξιδίων του αζότου. Γιατί τα θέματα αυτά συνδέονται. Ε, αυτά τα όρια είναι πολύ ψηλότερα για τα αυτοκίνητα που κινούνται με πετρέλαιο από ότι για αυτά που κινούνται με βενζίνη. Γιατί λοιπόν αυτά να επιτρέπεται να μολύνουν περισσότερο. Ε, εμείς έχουμε την ευκαιρία στο Ευρωκοινοβούλιο να αντιμετωπίσουμε και να βελτιώσουμε τον μολυσμένο αέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει τεχνολογία και η νομοθεσία θα πρέπει να ανταμείβει εκείνους τους κατασκευαστές αυτοκινήτων που κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση της υπάρχουσας τεχνολογίας. Πρέπει να έχουμε αυστηρότερους ε, ε, εξοπλισμούς δοκιμής για δοκιμασίες για να εξασφαλίσουμε ότι τα στάνταρα αυτά θα τηρούνται και στους δρόμους θα πρέπει να γίνει σοβαρή συζήτηση για το κατά πόσο χρειάζονται καν οι παράγοντες συμμόρφωσης εφόσον μπορούν να γίνουν μετρήσεις με ακρίβεια ε, μέσω των καλύτερων διαθέσιμων εξοπλισμών δοκιμών. Θα πρέπει λοιπόν τα αυτοκίνητα να δοκιμαστούν υπό κάθε πιθανή ε, περίσταση ε, και, αντί και καλύτερα έτσι, να μην βασιζόμαστε σε παράγοντες συμμόρφωσης. Δεν μπορούμε να έχουμε πλέον δικαιολογίες ότι δηλαδή δήθεν ε, α, κάτι τέτοιο θα βλάψει την υγεία των πολιτών τα στάνταρα που έχουμε λοιπόν επί χάρτου θα πρέπει να ισχύουν και στην πράξη, στον πραγματικό ο κόσμο, προ όφελο των ε, συμπολιτών μας. Για το Ρινιού, η Σουζάννα Σόρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσίασή του. Είναι σαφές ότι πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ πιο φιλόδοξοι όσον αφορά την μείωση των οξυδίων του αζότου από τα αυτοκίνητα, αν θέλουμε να τηρήσουμε τις μέσει μα περιβαλλοντικές. Αυτό όμω θα πρέπει να γίνει με βάση διαφορετική νομοθετική πρόταση από τη σημερινή. Ε, και μάλιστα αυτή με ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, με ένα ε, μελέτη αντικτύπου και με συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν νομίζω πως θα πρέπει να συζητήσουμε καν αυτήν το νομοθέτημα γιατί κάτι τέτοιο θα καθυστερούσε αυτή τη διαδικασία και θα δημιουργούσε βεβαιότητα για την αυτοκινητοβιομηχανία και για τα εκατομμύρια θέσεων απασχόληση που εξαρτώνται από την αυτοκινητοβιομηχανία. Εγώ λοιπόν είμαι υπέρ του να προχωρήσουμε εδώ γρήγορα ώστε και το Κοινοβούλιο να δείξει σαφή δέσμευση ώστε να μειωθούν ε, σημαντικά οι εκπομπές οξυδίων του αζώτου στο επόμενο ευρώ 6 ή και στο ευρώ 7 ε, και να απαλλαγούμε από τους παράγοντες συμμόρφωσης. Και θέλω να κάνω και μια σχετική ερώτηση προς την Επιτροπή, γιατί θα ήθελα να γνωρίζω γιατί σε αυτή την πρόταση τη σημερινή ο παράγοντας της συμμόρφωσης παρουσιάζεται μόνο με ένα μόνο αριθμό, χωρίς να γίνεται διάκριση για το περιθώριο σφάλματος, όπως είχε γίνει στην προηγούμενη νομοθεσία του 2015, που ήταν χωριστά αυτά τα δύο. Θα πρέπει λοιπόν να ξεχωριστούν οι ευθύνε που φέρουν οι κατασκευαστές των αυτοκινήτων, που είναι υπεύθυνοι για την τήρηση αυτού του ορίου 80 μιλιγκράμμ ανά... Ε, χιλιόμετρο. Ε, αυτό είναι το όριο, και, αλλά και να μοιραστούν την υπόλοιπη ευθύνη οι κατασκευαστές των εξοπλισμών ελέγχων και δοκιμών. Γιατί λοιπόν παρουσιάζεται έτσι όλο σαν ένα πράγμα και έπειτα. Ε, μιλάμε για το ότι υπάρχει μια έρευνα του Κοινού Κέντρου Ερευνών και ότι αυτή λέει πως μπορεί να μειωθεί αυτό το, το ε, περιθώριο ε, σφάλματος στο 0,32 πότε επιτέλους θα δημοσιευθεί αυτή η μελέτη και γιατί καθυστερεί τόσο, γιατί είναι σαφές ότι αυτό το περιθώριο σφάλματος, εφόσον πρέπει να αναθεωρηθεί προς τα κάτω, πρέπει να αναθεωρηθεί ε, και να γίνεται αυτό τακτικά, περιοδικά και ετησίω. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν επιστημονικά και τεχνολογικά στοιχεία, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να, πούμε, ε, να, να μιλήσουμε με βάσιμα στοιχεία. Ευχαριστώ και θα ήθελα να απαντήσεις σε αυτές μου τις ερωτήσεις. Πράσινη, Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομο, γιατί η Έστερ Λάγκη το είπε ήδη, ακούγεται τεχνικό το ζήτημα, αλλά είναι εξαιρετικά πολιτική φύση, γιατί αλλάζουμε τα στάνταρ που έχουμε συμφωνήσει στον κανονισμό του 2007. Το 2007 συμφωνήσαμε για στάνταρ τα οποία εκφράζονται στο άρθρο 5 για αυτοκίνητα σε πραγματικέ και κανονικέ συνθήκε χρήση. Κανονικέ συνθήκε χρήση. Έκτοτε προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε τις δοκιμές, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν επιμένουμε στα πρότυπα που συμφωνήσαμε το 2007. Διαφορετικά, αυτό που κάνουμε τώρα είναι 11-12 χρόνια αργότερα, ενώ είπαμε ότι τα αυτοκίνητα πρέπει να φτάσουν σε αυτά τα στάνταρ, πρέπει να μείνουν κάτω από αυτά τα στάνταρ, τώρα θέλουμε ε, λόγω των νέων δοκιμών, των νέων ελέγχων, να τους δώσουμε περισσότερη δυνατότητα να ρηπαίνουν. Και για όλους τους συναδέλφους που πάντοτε ζητούν ε, ε, την ουδετερότητα της τεχνολογίας, ας πούμε απαντήσετε γιατί σε αυτόν τον κανονισμό η, το πετρέλαιο επιτρέπεται να ρηπαίνει περισσότερο από ότι η βενζίνη. Για ποια τεχνολο... ουδετερότητα της τεχνολογίας μου μιλάτε τότε και επιπλέον θέλουμε να επιτρέψουμε στα αυτοκίνητα να ρηπαίνουν περισσότερο από ό,τι συμφωνήσαμε το 2007. Αυτό κάνουμε. Μπορεί να το λέμε περιθώριο σφάλματο, μπορεί να το λέμε παράγοντα συμμόρφωσης, αλλά αυτό που κάνουμε είναι ότι ε, μειώνουμε μια προδιαγραφή που συμφωνήσαμε το 2007 με το σαθρό επιχείρημα ότι δήθεν η έλεγχη δεν είναι επαρκή. Μα ήδη το 2007 είχαμε πει ότι το πρότυπο αυτό ισχύει για τα οχήματα υποκανονικέ συνθήκε χρήση. Εφόσον ο έλεγχο έλεγχος μιλά για περιθώριο σφάλματος και έχει πάντα περιθώριο σφάλματος, μα αυτό λέμε. Τα στάνταρ στη ΣΥΠΑ, τα στάνταρ στην Κίνα είναι χαμηλότερα. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων δουλεύουν γι' αυτό λοιπόν, για χαμηλότερες παιδιαγραφές. Η Ευρώπη λοιπόν δεν πρέπει να, να απογοητεύσει τους πολίτες της. Δεν θα πρέπει να γίνει αυτό με κατοξιδότηση πράξη. Είναι αλλαγή νόμου ε, ε, για ένα βασικό στάνταρ, μια βασική προδιαγραφή που συμφωνήσαμε το 7 και η Κομισιόν πάλι προσπαθεί να το περιορίσει από μόνη της. Και εμεί θα αντισταθούμε. Δεν έχω τώρα ομιλητή, λέει ο πρόεδρο για την ID. Α, συγγνώμη, ναι, είστε εδώ. Καταρχάς ευχαριστώ για την παρουσίαση από την πλευρά της Κομισιόν και τη συγκήτρια. Δεν είναι τώρα η ώρα να κάνουμε λογική συζήτηση. Το θέμα είναι να δούμε νομικός το πρόβλημα. Θέλω να επικεντρωθώ σε τρεις πτυχές. Πότε, οπότε συζητούμε εδώ, μιλούμε για μια νομική πράξη η οποία έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να το πω αυτό. Δηλαδή, αν τώρα το κοινοβούλιο θέλει να γελοποιηθεί τελείω, εντάξει. Τι να πω. Τώρα λέμε ξαφνικά θέλουμε να το αλλάξουμε. Ε, Φέτο το κοινοβούλιο αποφασίζει το Α και το χρόνο θα αποφασίσει το Β. Ε, μιλάμε και για νομική ασφάλεια. Ασφάλεια δικαίου. Και σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου του Φεβρουαρίου του 2020 που θα αρχίσει να ισχύει, λέγεται ότι η νομική πράξη ε, αποφασίζεται σε μια έκτακτη ε, διαδικασία και όχι σε, στη συνήθη διαδικασία. Θέλουμε με αυτή τη ε, διαδικασία να, κάνουμε, να καταστήσουμε υπεύθυνη την αυτοκινητοβιομηχανία επειδή δεν ε, έχει για την ασφαλή δικαίου και πρέπει να διρίξουμε και μια ματιά στην, στον συντελεστή για τις στατιστικά στοιχεία, για τις ε, ανακρίβειες που υπάρχουν σε διαφορά τις μετρήσεις, στατιστικά, γιατί κάθε τεστ, και έτσι που μου το εξήγησαν, κάθε τεστ γίνεται διαφορετικά. Και γι' αυτό δεν υπάρχουν πάντα συγκρίσιμα στοιχεία. Και απ' την άλλη, το, η συσκευή που υπάρχει στο αυτοκίνητρο αλλάζει σε σχέση με τις τιμές που καταγράφει. Και έχουμε και τις ανακρίβειες ε, τις τεχνικές. Οτιδήποτε και αν μετράτε κάθε φορά, πάντα θα έχετε να κάνετε μια ανακρίβεια, η οποία προκύπτει από την ίδια τη συσκευή μέτρησης. Οπότε έχουμε αποφασίσει κάτι, αλλά είμαστε ρεαλιστές, γιατί υποθετικά πάντα θα μπορούσε να υπάρχει μια συνέπεια, μια διαφορά μεταξύ αυτών που ε, μετρά κανείς σε ένα ε, εργαστήριο υπό τελείως πλασματικές συνθήκες και σε ό,τι μετρίαται στις πραγματικές συνθήκες, στην κανονική χρήση των οχημάτων. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας πάντα. Ευχαριστώ. Thank you for ECR, Ευχαριστώ για την ECR, η κυρία Ζαλιώσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε νομίζω ότι όλοι τα ίδια λέμε. Όλοι θέλουμε να προχωρήσουμε έτσι ώστε και οι πολίτες και οι κατασκευαστές να ξέρουν τι γίνεται σε ό,τι αφορά τον κανονισμό του 2007 και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί. Πρέπει να είμαστε έτοιμη μέχρι το τέλος του 2020. Κατά πάσα πιθανότητα και σύμφωνα με όσα μας λέει η Κομισιόν δεν θα είμαστε. Άρα αυτό τι σημαίνει, ότι ο κανονισμός του 2007 ισχύει, χωρίς τον παράγοντα της συμμόρφωσης. Και μάλλον από ό,τι φαίνεται η Επιτροπή που ψάχνει να βρει μια λύση δεν είναι έτοιμη. Θα ήθελα να μάθω από πού προκύπτουν αυτά τα νούμερα. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε τεχνικές απαντήσεις για να καταλάβουμε λίγο τη μεθοδολογία σύμφωνα με την οποία έγινε η έρευνα. Και το επόμενο ερώτημα είναι το εξή. Είναι έτοιμοι οι αυτοκινητοκατασκευαστέ, ε, έχετε μιλήσει με όλου. Και επίση, άλλο ένα ερώτημα. Όταν ε, κάναμε την ε, διαβούλευση στην Πολωνία στο άρθρο 11 Εμεί έχουμε πρόβλημα με το άρθρο 11 γιατί μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαιρούνται από την αγορά γιατί έχουν ε, εξοπλισμό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Αυτό εμείς θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερος ε, επικίνδυνο και θα υποβάλουμε σχετική τροπολογία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Κανιάτσινα, ε, σκιώδη συγγήτρια από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι μας ξέρουμε τι έγινε και ξέρουμε ότι πρέπει να διορθώσουμε αυτό που έγινε. Και χτες να είχαμε αναλάβει δράση, πάλι αργά θα ήταν. Υπάρχει νομική ανασφάλεια σε σχέση με τα όρια που πρέπει να πληρώνουν τα οχήματα και δεδομένου και του περιορισμένου χρονικού διαστήματος για να γίνουν τροποποιήσεις, εγώ προτείνω να εγκρίνουμε την πρόταση της Κομισιόν χωρίς τροποποίηση. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια α, ε, διαδικασία για την έγκριση τύπου για τα αυτοκίνητα, όχι μόνο για, τους αυτοκ... για την αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και για τους πολίτες. Ξέρω ότι έχετε βαρεθεί να με ακούτε να το λέω, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι μιλάμε για μία περίοδο 7 χρόνων για να εφαρμοστούν όλα αυτά. Μια αλλαγή μέσα σε λίγους μήνες θα έχει τεράστια αντίκτυπο στην οικονομία, στην απασχόληση, στις θέσεις εργασίας, στην αυτοκινητομηχανία και στο περιβάλλον. Το 0,43 και ο σχετικός παράγοντας συμμόρφωσης βασίζεται στην τεχνική ανασφάλεια που προκύπτει από τη χρήση των φορητών συστημάτων, των PEMS με αλλαγές στην θερμοκρασία, στην υγρασία και άλλους τεχνικούς παράγοντες που επηρεάζουν. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε το ίδιο επίπεδο ακρίβειας όπως έχουμε σε ένα ε, εργαστήριο. Ποτέ δεν πρόκειται να καταφέρουμε να, δούμε, να βρούμε πώς μετρούμε σε πραγματικές συνθήκες πράγματα που μετριούνται σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον ενός εργαστηρίου το ερευνητικό κέντρο είναι ένας ανεξάρτητος φορέας που τονίζει το θέμα αυτό. Δεν είναι οι κατασκευαστές που θα, που θα παρέμβουν εδώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα λέει ότι αυτό το αναθεωρεί κάθε χρόνο. Όπως εξελίσσονται τα PEMS βεβαίως μπορεί να υπάρξουν και αλλαγές. Και επειδή υπάρχουν και υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη αυστηροποίηση των ορίων για τις εκπομπές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει νέες τιμές για το 2021. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να εισαγάγουμε νέα επιπλέον ανασφάλεια, ούτε θα πρέπει να τιμωρήσουμε τους ε, κατασκευαστές επειδή δεν μπορούν να μας δώσουν πιο, ακριβή, ε, πιο ακριβείς συσκευές μέτρησης. και δεν θα πρέπει να κάνουμε κάτι που μακροπρόθεσμα θα μας κοστίσει και οικονομικά και κοινωνικά. Παρόλο που μπορεί σήμερα να φαίνεται πολύ ελκυστικό. Ευχαριστώ. Ωραία. Ε, Ευθείε ερωτήσει λοιπόν προ την Κομισιόν. Δύο λεπτά για τι απαντήσει σα. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Θα ξεκινήσω με το σχόλιο της εισηγήτριας που ανέφεραν και διάφοροι άλλοι βουλευτές, που είναι η δουλειά που κάνει το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο για τις πιθανή αλλαγή στην τιμή του περιθωρίου σφάλματος. Αυτό μπορούμε να πούμε σήμερα το τελευταίο στάδιο, προβλέπεται ε, ε, για την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου. Οι συνάδελφοι στο Κοινό Ερευνητικό Κέντρο θα χρειαστεί ακόμα 2-3 εβδομάδες για την ανάλυση των στοιχείων και έτσι θα φτάσουμε στο τέλος του έτου σίγουρα δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένη ημερομηνία. Σίγουρα η αναθεώρηση λοιπόν θα γίνει μετά ε, και αυτή είναι μια από τις αλλαγές που έχει εισάγει το Συμβούλιο και φυσικά το υποστηρίζουμε. Επίσης, σε σχέση με το γιατί έχουμε μία τιμή και γιατί δεν δίνουμε ε, περιθώριο ε, σφάλματος, αυτό ήδη έχει αλλάξει στο Συμβούλιο. Είναι καλή τροπολογία που επιφέρει σαφήνεια για το Ε, πώς ε, θα γίνει η αλλαγή της τιμής αυτής είναι καλή πρόταση για τη πιο τεχνική επεξήγηση της δουλειάς που κάνει το ερευνητικό κέντρο. Αυτό που μπορώ να σας προσφέρω σε αυτό το στάδιο είναι μια παρουσίαση που κάνουν οι συνάδελφοι από το κοινό ερευνητικό κέντρο και που επιθυμούν, είναι πρόθυμοι να έρθουν εδώ και να σας εξηγήσουν ακριβώς πώς προχώρησαν για τη μέτρηση του νέου πιθανού περιθωρίου. Σήμερα λοιπόν ε, εργάζονται ε, μάλλον έχουν ήδη εξετάσει το 70% του εξοπλισμού που υπάρχει στην αγορά, προχωρούμε προς 90%, δηλαδή τα αποτελέσματα είναι πολύ αξιόπιστα και πολύ στέρεα. Μπορούν λοιπόν να έρθουν οι συνάδελφοι εδώ να σας εξηγήσουν ακριβώς πώς προχώρησαν σε αυτόν τον έλεγχο. Τώρα, για το θέμα του κατά πόσο οι κατασκευαστές των αυτοκινήτων είναι έτοιμοι να το δεχτούν ή να το μειώσουν ή να δεχτούν τη μείωση. Ναι, είναι έτοιμοι. Πρόκειται για ένα περιθώριο το οποίο είναι εφικτό από ό,τι έχουμε καταλάβει και από ό,τι έχουμε δει σήμερα. Φαίνεται να είναι ενδιαφέρουσα ενδιαφέρον ε, και μπορεί να επιτύχει αποτελέσματα. Τώρα, για το Euro 7, σημαντική παρατήρηση είναι ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει τη δουλειά πάνω σε αυτό το project. Θέλουμε να κάνουμε την δεύτερη μελέτη στις αρχές του επόμενου έτους και την μελέτη αντικτύπου. Είναι η τελευταία μας εργασία γιατί εκεί ε, συνδυάζουμε ε, τα στοιχεία και είμαστε έτοιμοι να εισάγουμε αλλαγές όχι μόνο στα όρια, αλλά να υπάρξει συνοχή σε όλες τις κατηγορίες, να έχουμε όμως ένα ε, μελέτη αντικτύπου μέσα στο 2020 και να κάνουμε σχέδιο πρότασης το 2021 με την προϋπόθεση βέβαια ότι κάτι, αυτό θα πρέπει να εγκριθεί από τη νέα Επιτροπή. Η τεχνική δουλειά γίνεται από τις υπηρεσίες μας αλλά θα πρέπει να περιμένουμε για επίσημη έγκριση. Τώρα για τα όρια ε, εκπομπών για τα ε, πετρελοκίνητα και τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Αυτό είναι κάτι που οι νομοθέτες θα πρέπει να το σκεφτούν και θα πρέπει με τα πρότυπα Euro 7 να είμαστε βέβαιοι ότι θα ισχύσει η ουδετερότητα της τεχνολογίας. Νομίζω αυτά ήταν τα ερωτήματα. όχι, όχι. Ε, είπατε κάτι για το πόσο χρόνο έχουμε για να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το σχέδιο νομοθεσίας. έχει πει λοιπόν το δικαστήριο, ότι η περίοδος επεξεργασίας νέων προδιαγραφών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία επί της οποίας ισχύει αυτή η απόφαση. Η απόφαση αυτή δεν ισχύει γιατί έχει ε, υποβληθεί έφεση. Άρα έχουμε χρόνο περισσότερο μπροστά μας, ίσως θα μην το γνωρίζατε, αλλά έχουμε περισσότερο χρόνο. Ακόμα ένα σχόλιο όσον αφορά τις παράγοντες ε, συμμόρφωσης ε, ως ε, δικαιολογία για να μην ακολουθήσουμε αυτά που ισχύουν. Το, το δικαστήριο δεν αμφισβήτησε την φύση των παραγόντων ε, ε, συμμόρφωσης. Αυτή την απόφαση την έχετε ενώπιόν σας. Εσείς και το Συμβούλιο μπορείτε τώρα να αποφασίσετε αν θα διατηρήσετε αυτούς τους παράγοντες συμμόρφωσης ή όχι. Σας ευχαριστώ πολύ. Η εισηγήτρια τώρα έχει τον τελευταίο λόγο. Εγώ ήθελα να ελέγξω αν έχουμε ήδη αν ξέρουμε, έχουμε ήδη πει ότι με τους ε, σκιώδεις θα κάνουμε μια τεχνική συζήτηση με την Κομισιόν και το Κοινό Κέντρο Ερευνών στις 4 ε, Δεκεμβρίου. Επί τη βάση της σημερινής συζήτησης, ιδιαίτερα όσον αφορά τα τεχνικά ζητήματα, είναι καλό που έχουμε ήδη προβλέψει συνεδρίαση με, με το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο, ώστε να εξετάσουμε και να τους υποβάλουμε όλα αυτά τα ερωτήματα. Αυτό που θέλω να πω είναι καταρχάς ευχαριστώ για τις συμβολές σας, πολύ χρήσιμα τα σχόλιά σας και βέβαια όλη μας η Επιτροπή είναι δεσμευμένη να κάνει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια εφόσον μιλάμε για την ποιότητα του αέρα για τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Να συγκρίνω όμως αυτό που κάνουμε εδώ με αυτό που κάνουμε για τα πρόστιμα ταχύτητας. Ξέρετε πόσο μεγάλη προσοχή δέχτηκε αυτό το θέμα. Όλοι γνωρίζουμε πως αν πάρουμε ένα πρόστιμο, η αστυνομία σου λέει «Ναι, αλλά έτρεχες με 130 σε μία... σε ένα δρόμο που το όριο ταχύτητας ήταν 120 ε, ας πούμε, αλλά σου μειώνουν κατά 8 χιλιόμετρα την ταχύτητα την οποία κατέγραψε το ραντάρ. Γιατί υπάρχει ένα περιθώριο σφάλματος πάντοτε. Υπάρχει μια κάποια βεβαιότητα και οι κλίμακες... Δεν, ακόμα και οι, και οι ζυγαριές που έχουμε στο μπάνιο μας δεν είναι 100% ακριβίας ή εκείνες οι ζυγαρίτσες που χρησιμοποιούμε στην κουζίνα μας για να μετράμε τα μικροσκοπικά ποσά από τα υλικά που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε ένα γλυκό. Και γι' αυτό το πράγμα μιλάμε, συνάδελφοι, και πιέζουμε την Κομισιόν για το Euro 7 και εκεί αυτή είναι η βάση για τα όρια για τα αυτοκίνητα. Μιλάμε για εξοπλισμούς μετρήσεων και θα πρέπει να τα κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Um, Ευχαριστούμε. Το σχέδιο θα είναι για τον Ιανουάριο, αλλά επειδή είναι πολύ σημαντικό μπορεί να συμφωνήσουμε ότι αν εσείς με τους συντονιστές θέλετε άλλη μια συνάντηση ώστε να μην έχουμε μόνο συνάντηση μεταξύ ε, σχεδόν, αλλά να το συζητήσουμε όλοι μαζί, μπορούμε. Μην ανησυχείτε, μην ανησυχείτε. Θα είμαι έτοιμη. Ωραία, δεν ανησυχώ. Το Μάρτιο της επόμενης χρονιάς θα ψηφίσουμε εδώ. Ωραία, περνάμε στους συντονιστές τώρα.